Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε, παρακαλώ. Πριν να Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, Χθε είχαμε τη δυστυχή επέτειο των επιθέσεων στις Βρυξέλλες και χθε, ένα χρόνο ακριβώς μετά, στο Λονδίνο ε, έλαβε χώρα μια τραγωδία και θέλουμε να εκφράσουμε εκ μέρους της Επιτροπής μας όλη μας την υποστήριξη προς το Βρετανικό λαό ε, θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας ε, στα θύματα και στους συγγενείς τους και για να μην ξεχνάμε και να δείχνουμε αλληλεγγύη εμείς ως Ευρωπαίοι θα σας ζητήσω να σηκωθούμε όρθια και να τηρήσουμε ένας λεπτός Je vous annonce que Σας ανακοινώνω ότι οι αποφάσεις ε, που έλαβαν οι συντονιστές ε, στην χθεσινοβράδινη συνεδρίασή μας ε, έχουν τυπωθεί σε αντίγραφα τα οποία σας έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις μέχρι τις 12.30 θα θεωρήσουμε ότι οι αποφάσεις έχουν εγκριθεί. Ας ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Να δοκιμάσουμε πρώτα τις ε, κάρτες ψηφοφορίας και ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν ε, ε, έχουμε το σωστό αριθμό για την απαρτία. Η πράσινη είναι ένας παραπάνω, οπότε δεν θα ψηφίσω εγώ. Ωραία. Είμαστε σωστά. Ξεκινάμε. ξεκινάμε. Ξεκινάμε την ψηφοφορία για τις δεσμευτικές αιτήσει μειώσεις των εκπομπών αριών του θερμοκηπίου από τα κράτη-μέλη από το 2021 στο 2030 σχέδιο γνωμοδότησης με συντάκτρια την κυρία Κιλένεν. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται νομίζω, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Το ΕΛΚ έχει μία παραπανίσια ψήφου. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Λοιπόν, τώρα είναι σωστό, μου λένε. Να το προβάλλουμε στην οθόνη. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Κύριε Βέρνερ, φεύγετε στο επανειδήν. Δεν μας άκουσε. Γεια σας, στο επανειδήν. Συμβεβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Τμήμα 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, συμβαστική 6 έχει εγκριθεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. 62 απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές η 63 απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Μισό λεπτάκι μου λένε ότι η 66 έχει ήδη εγκριθεί. Διότι εγκρίθηκε η 64. Οπότε καταπίπτει. Και το ίδιο ισχύει και για την 42. Περνάμε λοιπόν στις ε, ταυτόσιμες τροπολογίες 67 και 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι 67 και 68 απορρίπτονται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. κατά αποχές 69 απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές 72 απορρίπτεται τροπολογία 70 υπέρ κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Γιατί είναι 70. Τέλος ψηφοφορίας. 19-19. Με μία αποχή απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Vous voulez le compromis 7. Να ελέγ... Θέλετε να ελέγξουμε τη συμβαστική 7. Ξεκινάει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 7... για τη συμβαστική 7. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Να μου έχετε εμπιστοσύνη κύριε Βίμπραντ. Ε, κύριε Βίμπραντ Κάμπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 80 απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 79 εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 81 απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές η 82 απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές η 83 εγκρίνεται η 84 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 84 ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας Η 84 δεν εγκρίνεται. 85 και 86 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές. Οι 85 και 86 απορρίπτονται. 100 Δεν ψηφίζουμε την 115, συνεχίζουμε παρακάτω. καταπίπτει αυτόματα ουσιαστικά. Θα, θα τα βρούμε μετά, λέει η Πρόεδρο. Συνεχίζουμε. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές η 88 απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ωραία σε ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Καλά κάναμε και ελέγξαμε διότι εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 90 υπέρ. Α, καταπίπτει 90, συγγνώμη. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 116 καταπίπτει επίση, διότι 87 δεν εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. 92 απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. 93 απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές 94 απορρίπτεται τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές η 95 εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές 96 απορρίπτεται η 97 υπέρ κατά αποχές η 96 λέει αλλά 97 ενώσε απορρίπτεται 9 ε, συμβιβαστική κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να ελέγξουμε αν θέλετε Oui, alors on ouvre le, le vote. Vous me regardez, euh, Monsieur Vimbonde de Camp. Τι λέτε κύριε Βαντεκάμπ. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική 9 πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Δώδεκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 12 απορρίπτεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές η 100 απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές να ψηφίσουμε ξεκινάει η ψηφοφορία για την 101 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται νομίζω αλλά να το ελέγξουμε ξεκινάει η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας η συμβαστική 10 απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην... τροπολογίε μία προ μία. Η 13 υπέρ. Κατά. αποχέ, Η 13 απορρίπτεται. Η 103 υπέρ. Κατά. αποχέ. Η 103 απορρίπτεται. 117. υπέρ, κατά, Λοιπόν, περιμένετε, λέει ο πρόεδρος. L'amendement 117 n'est pas... Η 117 δεν πρέπει να ψηφιστεί διότι 103 απορρίφθηκε. Περνάμε λοιπόν στην 104 υπέρ κατά αποχές 104 εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές 105 εγκρίνεται Τροπολογία 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 106 δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβιβαστική 11 εγκρίνεται. Συνεχίζουμε τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 15 εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 113 απορρίπτεται. Τροπολογία 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 114 απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 18 εγκρίνεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας ψηφοφορίας. Έχετε δίκιο κύριε Βαντεκάμπ, η 18 πράγματι απορρίπτεται. Η 19, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, το πρώτο τμήμα απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβιβαστική 1 εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές η τροπολογία 24 απορρίπτεται. Τροπολογία 27 και 28 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και οι δύο λοιπόν απορρίπτονται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά αποχές 26 απορρίπτεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές 29 απορρίπτεται τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ανοίγουμε την ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 32 απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 31 εγκρίθηκε. Η 3 υπέρ. Κατά. Να το επαναλάβουμε γιατί δεν είναι σαφές. Ποιος είναι υπέρ της 3. Μπράβο, καλύτερα έτσι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η συμβαστική 2 εγκρίνεται. Η 3 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 36 εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Μου ζητάνε επαλήθευση της 36. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λοιπόν η 36. Ήταν ε, ισοπαλία ουσιαστικά. Ε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 37 απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές 39 απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 5 δεν εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 40 δεν εγκρίνεται. 41 υπέρ. 40, κατά, συγγνώμη. Αποχές. Η 41 απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Η 6 εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 43 απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 45 απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές η 44 εγκρίνεται τραπολογία 22 υπέρ κατά αποχές 22 εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ Ε, λοιπόν, να επαληθεύσουμε την 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 εγκρίνεται. Να μου έχετε εμπιστοσύνη κύριε Βαντεκάμπ. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 23 κανονικά απορρίπτεται αλλά να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Μάλιστα καλά κάναμε που επαληθεύσαμε. Και ψηφίζουμε επί του συνόλου της γραμμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή, η έκθεση, γνωμοδότηση ε, γκρίνεται και ε, ευχαριστούμε κυρία Κελέναν. Και συνεχίζουμε. Nous continuons par le vote Συνεχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία για την παράσταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Η συγκήτρια κυρία Αγιάλα Σάντερ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλιστα, άρχεται ψηφοφορία για την 72 δεύτερο μέρος, έτσι. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές οπότε να το επαληθεύσουμε. Ε, πέρας, ε, ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας. Α, ήταν πολύ σαφή τα πράγματα τελικά. Αλλά δεν σηκώνεται το χέρι, γι' αυτό. Και εγώ τα μάτια μου τα έχω στα νύχτα. Και δεν είναι καν δέκα. Η τροπολογία 75 απορρίπτεται. Η τροπολογία 76. Η τροπολογία 75 εγκρίνεται, συγγνώμη. Η 76 Λοιπόν, εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ο συμβασμός 2 και τώρα περνάμε στην τροπολογία, στην τροπολογία 91 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφή τα πράγματα, Οπότε ψηφίζουμε επί του 91. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία 91 ε, δεν, απο, δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Α, θέλετε να, ελέγξουμε το 95. Εντάξει. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, η τροπολογία 95 δεν εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 18, ε, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στο συμβασμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. προφορική τροπολογία του κυρίου Ζήλε. Θέλετε να μας παρουσιάσετε κύριε Ζήλε. Όχι. Α, ναι. Ναι, όπως βλέπετε, θέλω να προσθεθεί και το ελεγκτικό σενέδριο στο κείμενο και στην τροπολογία. Y a-t-il Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτήν την προφορική τροπολογία. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις βουλευτές για να μην γίνει αποδεκτή η προφορική τροπολογία. Nous avons assez de députés. Nous avons assez de députés. Cet amendement aura. Αυτή η προφορική τροπολογία λοιπόν δεν θα τεθεί προς ψήφιση. Και συνεχίζουμε. Τροπολογία 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες Δεν εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ, κατά,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 32 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφή τα πράγματα άρχιτη ψηφοφορία η εντροπολογία 32 πέρας ψηφοφορίας η τροπολογία 32 δεν εγκρίνεται περνάμε στο συμβασμό 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβασμό 45. Ε, τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 55 καταπίπτει Ναι, σας ακούω κύριε Πίπερ. Δεν ξέρω αν ε, κατάλαβα σωστά, στην τροπολογία 54, την, την εγκρίναμε μάλλον, και στη συνέχεια ψηφίσαμε και για την τροπολογία 2. Μα η 54 ε, εγκρίθηκε. Ναι, η 54 εγκρίθηκε. Είμαι βέβαιος, απολύτως βέβαιος, γι' αυτό που σας λέω a été rejeté. Il n'a pas été adopté. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε επανήθευση, έτσι. Διότι εγκρίθηκε. Ε, μάλλον απορρίφθηκε, δεν εγκρίθηκε. Δεν μπορούμε όμω να πάμε τρει ψήφου, τρει ψηφοφορίε πίσω κάθε φορά. Έτσι. Θέλετε επαλήθευση. L'avant-dernier, il y en avait trois, deux avant. Il y en avait deux avant, M. Riquet. Είχαν γίνει και ψηφοφορίες πριν. Λοιπόν, εντάξει, τροπολογία 54. Εντάξει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 54. Πέρας ψηφοφορίας. και απορρίπτεται. Το είχαμε πει ότι είχε απορριφθεί βέβαια. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, να παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται και καλά κάναμε και παληθεύσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στο συμβασμό 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται. Να το παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Η τροπολογία 67 όντως απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα περάσουμε με λειτουργική ψηφοφορία στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και προχωράμε. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και ο εισηγητής μας εξακολουθεί να είναι η κυρία Γιάλα Σάντερ. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές η 3 απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές η 6 απορρίπτεται περνάμε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές οι 2 εγκρίνεται Πάμε στην ε, τροπολογία 12. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα της 12 εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 13. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 14 εγκρίνεται τροπολογία. Λοιπόν, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία Η 14 εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 16 απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές η 17 εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές η 18 δεν εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές η 21 δεν εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές η 25 απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 3 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 4 συμβιβαστική. Δεν είναι σαφές. Ε, κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω ότι κανονικά δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 4 λοιπόν ψηφίζουμε. Εγώ νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, πράγματι εγκρίνεται η συμβιβαστική 4. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές. Η 5 εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές. Η συμβιβαστική 6 εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 39 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 7 εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 46 εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε επί του συνόλου του τελικού κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 2 κατά, δεν υπάρχουν αποχές. Η έγκριση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Et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 και συνεχίζουμε με το σημείο 17. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σημείο 17 το οποίο αφορά την εξέταση και την παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Κόλσον. Καλημέρα και καλώς ορίσατε για 10 λεπτά περίπου για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού 181 του 11 που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν. Και θα του ζητήσω, αν έχει την καλοσύνη, να μας πει με λίγα λόγια περί τίνος πρόκειται αυτή η πρωτοβουλία της Κομισιόν για τα δικαιώματα των ε, επιβατών σε διατροπικές μεταφορές. Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι τις 25 Μαΐου. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να ακούσουμε και κάποιες εξηγήσει ε, από την Κομισιόν όσον αφορά τις προθέσεις της και το χρονοδιαγραμμά της. Η Επιτροπή Μεταφορών ε, επιθυμεί εύκολη και προσπελάσιμη ε, προσπελασμένες συγκοινωνίες ε, για τους ε, πολίτες και βάζουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ευκολία πρόσβασης για τους ανθρώπους μειωμένης κινητικότητας. Είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή μας. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός ε, του οποίου θα παρουσιάσω είναι ο τελευταίο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Έχει να συμπληρώσει του κανονισμού που έχουν να κάνουν με τι αερομεταφορέ, τι ε, μεταφορέ με τρένο και τι θαλάσσιε μεταφορέ. Όπω γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη περιοχή του κόσμου όπου οι επιβάτε έχουν δικαιώματα συγκρίσιμα διευρυμένα όποιο και να είναι το μέσο μεταφοράς. Μετά από δυόμιση χρόνια λειτουργίας του κανονισμού αυτού μπορούμε να πούμε, και είναι και το πιο βασικό συμπέρασμα αυτό θα έλεγα, ότι λειτουργεί καλά. Έχει γίνει αποδεκτό από τους μεταφορείς που το χρησιμοποιούν και για να ε, διαφημίσουν, να προωθήσουν το δικό τους τρόπο μεταφοράς, εφαρμόζουν τις σχετικές ε, διατάξεις και οι επιβάτε επίση κρίνουν θετικά τους κανόνες αυτούς. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ορίσει μια αρχή που ασχολείται με την εφαρμογή και έχουν ε, ψηφίσει και νόμο σχετικά με τις κυρώσει που μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων αυτού του νομοθετήματο. Οι κριτικές που θα μπορούσε κανεί να ε, ασκήσει δεν έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του κανονισμού, έχουν να κάνουν με κάποιες από τις διατάξεις του οι περισσότερες από διατάξεις του κανονισμού περιορίζονται στις υπηρεσίες, στις μεταφορές πάνω από 250 χιλιόμετρα. Ε, και αυτό το επικρίνουν οι ενώσεις καταναλωτών. Επίσης, τα κράτη-μέλη μπορούν να εξαιρέσουν τις αμυγός εθνικές υπηρεσίες έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2021 και 12 κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις εξαιρέσεις τουλάχιστον έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι από αυτούς θα επεκτείνουν αυτές τις παρεκκλήσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Δύο πάντως ε, ε, έχουν ήδη, το έχουν ήδη αναφέρει, ότι θα, έχουν αναφέρει θα το πράξουν. Είναι λοιπόν αυτά κάποια όρια στον κανονισμό. Το προβλέπουν όμως οι διατάξεις του. Ε, ο κανονισμός επιβάλλει στα κράτη-μέλη μόνο ε, την, ε, το να ορίσουν μία ε, υπηρεσία ε, που να χορηγεί υπηρεσίες στο άτομα με δικές ανάγκες, στο άτομα με αναπηρία, συγγνώμη. τώρα, αν κάποια, κάποιες χώρες έχουν βέβαια δώσει περισσότερα κέντρα, περισσότερους σταθμούς όπου μπορεί να υπάρξουν τις υπηρεσίες, έχει καλός, αλλά κάποιοι άλλοι επέλεξαν μόνο μία. Είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανησυχητικό. Κάποια κρατημέλη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις, αλλά κάποια άλλα όχι. Η νέα εκστρατεία ε, ενημέρωση της Κομισιόν επικεντρώνεται στα, κοινωνικά δίκτυα και αυτό, κοινωνικά μέσα δικτύωσης και αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο διότι όπως ξέρετε οι νέοι είναι αυτοί που κυρίως παίρνουν αυτά τα λεωφορεία που κάνουν μεγάλες διαδρομές, ε, επειδή είναι και πιο φτηνά. Μου στήσετε να πω δύο λόγια για την πρωτοβουλία που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών στις μεταφορές με συνδυασμένα μέσα. Ο οδικό χάρτη έχει δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο σχετικό και έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Βεβαίω είναι πολύ νωρί για να σα δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για αυτή την πρωτοβουλία. Οπότε οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν μετά και την αξιολόγηση αντικτύπου. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το στάδιο μπορούμε ήδη να ε, πούμε τα εξής. Καταρχήν, έχουμε όλο και πιο πολλές υπηρεσίες μεταφορών ε, συνδυασμένων που παρουσιάζονται ως συνδυασμένε μεταφορές μάλιστα, χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα μεταφοράς, διαφορετικά, διαδοχικά, από τον επιβάτη. Με ένα εισιτήριο γίνεται αυτό. Συνήθως αυτό αφορά ε, συνδυασμό αερομεταφορές τρένα. Ε, στην Γκάρτη Μιντή συμβαίνει αυτό ε, ας πούμε ή ε, Υπάρχουν όμως και άλλες, άλλες συνδυασμοί, πούλμαν φέρει, ε, σιδηρόδρομος ε, φέρει, πλοίο δηλαδή ε, και τα λοιπά. Θα αυξηθεί αυτή η τάση στο μέλλον. Οι κανονισμοί μας όμως έχουν σχεδιαστεί αναμέσω μεταφοράς. Δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτές τις νέες υπηρεσίες. Και αυτό βεβαίως είναι επιζήμιο για τους επιβάτες, ιδιαίτερα ε, όταν παραδείγματο χάρη χάσουν ε, την ε, αλλαγή από το ένα μέσο στο άλλο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δώσουμε στον επιβάτη τη δυνατότητα προσφυγής εφόσον ο ίδιος επιβάτης οργανώνει το ταξίδι του παίρνει λοιπόν δύο διαφορετικά μέσα μεταφοράς ξεχωριστά και η καθυστέρηση του ενός τον κάνει να χάνει το άλλο. Και υπάρχει και το θέμα των ε, επιβατών με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δύο αυτές περιπτώσεις. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα ξεκινήσει το 2018 μάλλον προς το τέλος του 2018 και όχι τόσο στην αρχή, δηλαδή του χρόνου. Αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στο μέλη που επιθυμούν να μιλήσουν. Μπάρτ, παρακαλώ. Κύριε Μπάρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Κολσόν, για την παρουσίαση. Θα συνεχίσω στα γερμανικά, γιατί σημειώσουμε είναι στα γερμανικά. Ε, ε, Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις εξηγήσει και για την έκθεση, η οποία δείχνει αναδεικνύει ορισμένα θέματα τα οποία χρήζουν της ε, προσοχής μας παρά το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος ε, μας είπε ότι η εφαρμογή του κανονισμού είναι ικανοποιητική. Λείπουν βεβαίως ορισμένα στοιχεία από τα, ε, από τα κράτη-μέλη για τις διασυνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των ε, στοιχείων. Φαίνεται για παράδειγμα από τις πληροφορίες που έχω ότι έχουν επιβληθεί λίγα πρόστιμα ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι και στις περιπτώσεις που ε, καταβάλλεται κάποια αποζημίωση ή έχει υποβληθεί κάποιο παράπονο, δεν υπάρχει υποχρέωση ο φορέας παροχής υπηρεσιών να καταχωρίζει ε, κάπου ε, το εκάστοτε περιστατικό. αντίστοιχα χαρακτηριστικά, αντίστοιχα λίγες είναι οι πληροφορίες έχουμε από τις περισσότερες χώρες Μόνο από την Ισπανία ε, έχουν ε, υποβληθεί 1.200 τέτοια περιστατικά. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για τις εξαιρέσεις του κανονισμού. Γιατί οι επιβάτες, οι πολίτες δεν μπορούν να κατανοήσουν επαρκώς και πλήρως για ποιο λόγο ε, δίνεται αυτή η δυνατότητα εξαίρεσης. Η ενημέρωση είναι το α και το ω ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις ακόμη. Πολλοί επιβάτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ε, στις αεροπορικές μεταφορές ή στους σιδηροδρόμους, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει ε, σε επαρκή βαθμό ε, για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ταχύτατα μια λύση όσον αφορά την πρόσβαση των ε, ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ε, στους ε, τερματικούς σταθμούς. Ακούστηκε ότι έχει, έχει τεθεί ένας στόχος να επιτευχθεί κάτι τέτοιο έως τα τέλη του 2018. Μου φαίνεται όμως ότι είναι πολύ αργά. Ακόμη και αυτός ο στόχος πρέπει να γίνει κάτι νωρίτερα. Επίσης, ε, όπως είπα, οι καταναλωτικές ε, οργανώσεις διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι υπάρχει ελλειπής πληροφόρηση ε, γύρω από τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, για το γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία στην υποβολή καταγγελιών και παραπώνων, ούτε υπάρχουν σε πολλές χώρες φορείς οι οποίοι να ε, διαχειρίζονται την, ε, τα περιστατικά διαφορών μεταξύ των εταιριών και των επιβατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήματα. Η Κομισιόν έχει πληροφορίες για τις χώρες οι οποίες δεν θα εφαρμόσουν ε, αυτά τα δικαιώματα έως τον Φεβρουάριο. Υπάρχουν κάποιες ε, εξελίξεις ε, σε αυτές τις χώρες έχουν ενδεχομένως προγραμματιστεί κάποιες ε, επενδύσεις, έχουν αναλυφθεί μέτρα. Είπατε επίσης ότι μπορεί να γίνει μια μεγαλύτερη πληροφόρηση των επιβατών μέσα των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει γίνει ήδη ή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιβάτες να γνωρίζουν όλες τις ε, απαραίτητες πληροφορίες προτού αποφασίσουν ποιον τρόπο μεταφοράς θα επιλέξουν. Ε, uh, κύριε Στυλίσκα, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, ε, θέλω να σας πω κατευθείαν ε, ότι μόλις τελειώσω τις ε, ερωτήσεις μου θα πρέπει να φύγω να πάω στην Επιτροπή Ήτρε. Όχι ότι δεν με ενδιαφέρουν, αλλά πρέπει, ε, υπάρχει μια σημαντική ψηφοφορία. Και ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Έχω διαβάσει μόνο την έκθεση, ε, πρέπει να σας πω. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου τον κανονισμό. δεν ξέρω λοιπόν αν αιτιολογείται το να πει κανεί οτι ότι μέχρι στιγμής μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν ζητήσει εξαίρεση, σαν να περιμένουμε ε, την 28η Φεβρουαρίου 2017 ε, ε, για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη που θα ζητήσουν εξαίρεση. Ε, ε, νομίζω ότι θα αρκούσε να πείτε ότι δύο είναι τα κράτη-μέλη που έχουν ζητήσει εξαίρεση για να μας πείτε σας παρακαλώ και ποια είναι αυτά τα δύο κράτη-μέλη. Δεύτερον, όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού, ας μην ξεχνούμε ότι το φθινόπωρο η Κομισιόν θα υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση που θα αφορά αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και τα συμπεράσματα που ακούσαμε σήμερα θα αντικατοπτρίζονται σε αυτή την νομοθετική πρόσωπο, πρόταση. Ε, ξέρω ότι ο, ο χαρακτήρας και η φύση αυτού του νομοθετήματος θα είναι διαφορετικό, αλλά παρόλα αυτά κάπως θα αντικατοπτρίζονται αυτά που ακούσαμε σήμερα εδώ. Τρίτον, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι μετακινούνται στην Ευρώπη και χρησιμοποιώ και εγώ λεωφορεία, ε, αλλά στους τερματικούς σταθμούς δεν βλέπω ποτέ ε, τις πληροφορίες που μπορεί κανείς να λάβει σε ένα αεροδρόμιο για παράδειγμα. Τι θα κάνει η Κομισιόν για αυτό το πρόβλημα. Και τέλος, μεταξύ των κρατών μελών που δέχονται τους μεγαλύτερους αριθμούς ε, παραπώνων, Ισπανία, Γερμανία, η δική μου χώρα, αυτό ε, ε, οφείλεται στο γεγονό ότι πράγματι γίνεται ε, παραβίαση των δικαιωμάτων των ε, επιβατών ή μήπως οφείλεται στο γεγονό ότι το σύστημα εκεί λειτουργεί καλά. Τι από τα δύο συμβαίνει. Και ποια η στάση της Κομισιόν απέναντι στα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτό το θέμα. Τη ε, μη υποβολή καταγγελιών λόγω τη μη καλή λειτουργία του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Κράμερ. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίαση αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω όμω γιατί η Κομισιόν δεν θεωρεί ότι ε, χρειάζεται αναθεώρηση αυτός ο κανονισμός. Διότι τα δικαιώματα των επιβατών στην πραγματικότητα των επιβατών Πούλμαν ε, ε, ενισχύουν τον ε, αθέμητο ανταγωνισμό ε, εναντίον του σιδηροδρόμου και των άλλων μορφών μεταφοράς. Δεν πληρώνουν τίποτα, δεν πληρώνουν διόδια τα, τα πούλμαν, σε αντίθεση με, το, με, τα, με τους σιδηροδρόμους. Επίσης, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, τα δικαιώματα αυτά εξασφαλίζονται στην περίπτωση του σιδηροδρόμου ε, από αποστάσεις 50 ε, χιλιόμετρων και πάνω. Ε, το αντίστοιχο ε, στα Πούλμαν είναι 250 χιλιόμετρα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Όταν ε, καταρτίστηκε και εκπονήθηκε ο κανονισμός αυτός, δεν είχαν διαδοθεί ακόμη τόσο πολύ τα πούλμα και τα λεωφορεία, τουλάχιστον στη δική μου χώρα. Αλλά πλέον έχουμε συλλέξει εμπειρία. Επίσης, βλέπω ότι δεν έχετε πληροφορίε. Ξέρετε σε τι οφείλεται αυτό. Στον κανονισμό για του σιδηροδρόμου αναφέρεται ότι η συνδρομική επιχείρηση δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της τον αριθμό και το είδος των ε, καταγγελιών που λαμβάνει ε, ε, τον χρόνο επεξεργασίας και την κατάληξη, το αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών αυτό στο σιδηρόδρομο. Αντίστοιχο, αντίστοιχη διάταξη δεν υπάρχει για τα πούλμαν. Γιατί δεν λέτε να υπάρχει και για τα ε, πούλμαν, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ε, να, να, υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Λέτε ότι δεν έχετε ε, αριθμό, ε, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των καταγγελιών. Μα πώ να τα έχετε, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση να καταχωρίζονται κάπου τα παράπονα αυτά, ούτε άλλα στοιχεία. Α γίνει αυτό και μετά θα, δούμε, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Βλέπω ότι σε σχέση με το 2015, Οι απολεστήσεις αποσκευές στα Πούλμαν αυξήθηκαν κατά 25%. Μα δεν σας ανησυχεί αυτό. Φανταστείτε κάτι τέτοιο να έχει γίνει στα αεροπλάνα ή στα, ή στα, ή στα τρένα. Θα έχει γίνει χαμός. Αλλά εδώ βλέπω ότι δεν σας ανησυχεί καθόλου κάτι τέτοιο. Ο αθέμητος ανταγωνισμός συνεχίζεται. Δεν γίνεται δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον αυτό που χρειαζόμαστε ε, θα ήταν να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ε, για τις απο, αποζημιώσεις είχαμε εξελίξει τα τελευταία χρόνια στους ιδεοδρόμους και στα αεροπλάνα. Γνωρίζετε για τις καθυστερήσεις άνω των 5 ώρων είχαμε πει εμείς. Το δικαστήριο όρισε το όριο αυτό στις 3 ώρες. Ε, ε, κάτι αντίστοιχο πρέπει να θεσπιστεί και για τα, για τα, για τα λεωφορεία. Όλες αυτές τις εμπειρίες που έχουμε, ε, που έχουμε συλλέξει τα τελευταία χρόνια ε, νομίζω ότι χρειάζεται να τις αξιοποιήσουμε και εδώ ο Τζος Μπαρ έχει δίκιο. Ε, χρειαζόμαστε ίσως όρο του ανταγωνισμού τουλάχιστον ως προς την υποχρέωση πληροφόρησης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Δεν έχω πολλά ερωτήματα γιατί τα περισσότερα που ήθελα να θέσω τέθηκαν. Θυμάμαι όμως ότι εγώ ήμουν η διαπραγματεύτρια τότε πριν από 10 χρόνια, ε, όχι 8, το 2009 πρέπει να ήταν όταν ε, ε, θεσπίστηκε αυτός ο κανονισμός. Ε, είναι πραγματικά απογοητευτικό. Ε, διότι ήταν η, η, πρώτη, το πρώτο νομοθέτημα για τα δικαιώματα των επιβατών των πούλμαν και των λεωφορείων και από αυτή την άποψη είναι απογοητευτικό το, το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ε, επιτευχθεί η πλήρης και ικανοποιητική εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Ε, και αυτά τα 250 χιλιόμετρα ε, θυμάμαι ότι ήταν μια συμβαστική στάση ε, γιατί υπήρχαν κράτη τα οποία ήθελαν ακόμα μεγαλύτερες αποστάσεις. Ο κύριος Τέλισκα ρώτησε ποιε είναι αυτές οι δύο χώρες που έχουν ζητήσει εξαίρεση. Επίσης γνωρίζαμε τότε ότι υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη που είχαν θεσπίσει ήδη εθνικά δικαιώματα επιβατών, κάποια που δεν, που δεν είχαν θεσπίσει κάτι αντίστοιχο. Ε, Ιδίω ε, ω προ εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν είχαν θεσπίσει δικαιώματα επιβατών, ε, ποια είναι η πορεία τη εξέλιξη τη εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Η κυρία Φώστερ, παρακαλώ. Thanks. Just a brief point, because I ε, δύο λόγια να πω, γιατί πολλοί από εμά και η κυρία Μάσνερ θα θυμάστε κάποιε από τι συζητήσει που είχαμε εδώ και κάποιε από τις προκλήσεις. Δεν νομίζω ότι γίνεται ε, οτιδήποτε σκεμμένα από οποιονδήποτε. Ε, ξέρετε και να το ρυθμίσουμε εμεί τα κράτη-μέλη πρέπει να ασφαλίσουν ότι θα το εφαρμόσουν ε, να, και ίσω να πρέπει να φτιάξουμε και άλλο κανονισμό γιατί δεν νομίζω θα επιτύχουμε τα αποτελέσματα με την εφαρμογή ε, αλλά θυμάμαι από του συναδέλφου που ήταν εδώ τότε. Ε, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανεί τη διαφορά μεταξύ ενός ταξιδιού με πούλμαν και σε ορισμένε χώρε τα ταξίδια με πούλμαν είναι μεγαλύτερα από τι άλλε, με λεωφορείο συγγνώμη ε, σε ε, σχέση με ένα πούλμαν ξέρετε όταν ένα λεωφορείο μένει κολλημένο στην κίνηση για ώρες και ώρες που συμβαίνει σε αυτοκινητοδρόμους ιδίως γύρω από πόλεις τότε η πρόκληση είναι το πώ λύνεται αυτό το ζήτημα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο αυτό που μα προτείνει η Κομισιόν σήμερα ε, και που συζητάμε αυτά τα θέματα. Και νομίζω θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και πρόβλημα να συλλέξετε πληροφορίε από ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά το ποια είναι τα προβλήματα και το τι έχει γίνει για να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά το πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, είναι οι επιβάτε μειωμένη κινητικότητα. Είπατε ότι χρειάζεται ακόμα πολύ μελέτη. Και ξέρετε, πιστεύω ότι αν έχετε κάτι συγκεκριμένο μπορείτε να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά ε, για μένα ευχαριστούμε που ήρθατε να μας κάνετε μια ενημέρωση, αλλά καλό θα ήταν να έρθετε να μας δώσετε και κάποιες απαντήσεις. Ε, όχι ότι κάποιο να μας πείτε δηλαδή ότι κάποιο θέλει κι άλλο ένα κανονισμό, απλά να μα πείτε περισσότερε απαντήσει για το πώ πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Foster. Je redonne la parole à Monsieur Colson. Ο κύριος Κόλσον τώρα για να απαντήσει στα ερωτήματα που σας έχουν απευθυνθεί. Oui, merci, Madame Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, το ζήτημα των κυρώσεων είναι κάτι που επανέρχεται διαρκώς στο τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών και γενικότερα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη έχουν τεράστιο περιθώριο λεγμών ε, όσον αφορά τα κείμενα που αποφασίζουμε, διότι το μόνο που τους επιβάλλουμε είναι να έχουν κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Αυτό λοιπόν επιτρέπει στα νομικά συστήματα των κρατών μελών τεράστιο περιθώριο ελιγμών, οπότε τεράστια ποικιλομορφία και εκεί είμαστε λίγο αδύναμοι εμείς. Προσπαθούσαμε να το δουλέψουμε λίγο στον τομέα των αέριων μεταφορών, αλλά δεν είναι εύκολο. Και αυτό εξηγεί το γεγονό οτι ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, πάνε και επιβάλλουν κυρώσει συστηματικά σε κάθε παραβίαση, ενώ άλλα, αντιθέτως, προτιμούν να έχουν μια πιο ολιστική προσέγγιση, να ε, βάζουν λιγότερα πρόστιμα, ίσως ε, ψηλότερα, για κάποια άλλα να μην ε, βάζουν χρηματικά πρόστιμα αλλά να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτό οδηγεί ε, στις τεράστιες διαφορέ που βλέπουμε στους πίνακες. Είναι δύσκολο να δράσει ε, συγκεκριμένα η Κομισιόν υπό τέτοιες συνθήκες. Η υπόθεση της Ισπανίας εξηγείται με δύο τρόπους. Πρώτον, οι μεταφορές με πούλμαν είναι τρομακτικά σημαντικές στην Ισπανία, περισσότερο από τις άλλα κράτη-μέλη. τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων εδώ και πολλά χρόνια. Δεύτερον, οι ελεγκτικές αρχές ε, όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού μερικές φορές έχουν ε, υπερβολικά πολλά καθήκοντα σε σχέση με τον κανονισμό. Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία. Αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια υποσημείωση ε, στην έκθεση αυτή. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται, οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην αρχή ε, σχετίζονται με τις κυρώσεις αυτές αλλά καλύπτουν μεγαλύτερο πεδίο από ότι ο κανονισμός. Έτσι εξηγείται ότι στην Ισπανία έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό καταγγελιών και κυρώσεων. Όσον αφορά το ζήτημα των εξαιρέσεων, είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι έχουμε εδώ ένα κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ πριν από δυόμιση χρόνια. Δεν είναι πολύ για να χρειάζεται να τροποποιήσουμε ένα κανονισμό αυτού του είδους. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη ότι θα είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία για αυτούς να αποφασίσουν αν θα παρατείνουν ε, τι εξαιρέσει για τις εθνικέ του υπηρεσίε ε, για περισσότερο χρόνο ή όχι προς το παρόν η Πορτογαλία και η Εστονία ε, το επεσήμαναν, υπάρχουν ίσως και άλλες, αλλά πρέπει να το αποφασίσουν σχετικά πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Ε, η τερματική σταθμή Πούλμαν ε, και λεωφορείων είναι σίγουρα ένα πρόβλημα, αλλά ο κανονισμός έχει εκπονηθεί έτσι που νομικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιβάλλουμε πάνω από ένα τέτοιο τερματικό σταθμό σε ένα κράτο μέλο. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την αποτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κάποια κρατημέλη έχουν ε, προχωρήσει περισσότερο από άλλα στον τομέα αυτών. Η εκστρατεία ενημέρωση τη Κομισιόν έχει ξεκινήσει και βασίζεται κυρίω στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτή η επιλογή έγινε. Και όπως είπαμε η επιλογή αυτή θα πρέπει να, έχει ε, να επηρεάσει τον ε, κανονισμό για τις οδικές μεταφορές γιατί όλο και περισσότερο ε, χρησιμοποιούν οι νέοι το πούλμαν ή το λεωφορείο αντί για το τρένο γιατί το θεωρούν πολύ ακριβό. Όλο και περισσότερο λοιπόν ταξιδεύουν με πούλμαν. Το θέμα αυτό λοιπόν της εκστρατείας ε, ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, θα πρέπει να φέρει κάποια αποτελέσματα. Οι πληροφορίες η Κομισιόν ε, έχει εκδώσει φυλάδια και αφήσει. Δεν τα βρίσκουμε παντού βέβαια και πάντα και ε, επίσης δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ε, να αναρτώνται στους σταθμούς των πούλμα λεωφορείων. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση τους, να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τα φυλάδια αυτά να μοιράζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα όσον αφορά τη διαφορά που ανέφερε και ο Κράμερ, η διαφορά μεταξύ του ζητήματος των εξαιρέσεων ε, για το Πούλμαν ε, και για τους σιδηροδρόμους. Πιστεύω ότι εκεί αναφερθήκατε κυρίως ε, στη γερμανική περίπτωση και στη Γερμανία πράγματι οι σιδηρόδρομοι δεν έχουν εξαιρέσεις. Γιατί, γιατί είναι επιλογή της γερμανικής κυβέρνησης. Αλλά αν δείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες, εκεί αντιθέτως οι σιδηροδρομικές μεταφορές περιλαμβάνουν πολύ περισσότερες εξαιρέσεις από ό,τι για τα πούλμαν. Η δυνατότητα που έχουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να εξαιρέσουν ε, ε, εθνικές ε, υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης χρησιμοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατάσταση λοιπόν των εξαιρέσεων, αν κάνουμε τη σύγκριση των δύο τρόπων μεταφοράς, δεν είναι και τόσο προβληματική ούτε ε, επιζημία για το πούλμαν όσο θα σκεφτόταν κανείς ε, υπέρ και υπέρ των σιδηροδρόμων. Και μάλιστα αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα εστιαστούμε για την αναθεώρηση του κανονισμού για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτά μέσα σε άκρες κύριε Πρόεδρε που αυτά ήθελα να πω για τις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Κύριε Κράμερ, έχετε μια παρατήρηση. Ε, σε, ένα σημείο δεν είχατε δίκιο. Τότε η Κομισιόν και ε, το Συμβούλιο ήθελαν να καταρτιστούν, να θεσπιστούν ε, δικαιώματα μόνο στις διεθνείς ε, μεταφορές. Και είχαμε πει τότε ότι είναι παράλογο αν κάνω ένα ε, ταξίδι από τη μία χώρα στην άλλη να ισχύουν ορισμένα δικαιώματα ενώ αν, το κάνω εντός της ίδιας χώρας τότε δεν έχω δικαιώματα. Είχαμε διαπραγματευτεί μέχρι τότε ε, έως τις ε, μέχρι τις 3 ώρα τη νύχτα. Γι' αυτό και η Γερμανία ε, ορθώς τότε είχε τηρήσει τη στάση και, είχαμε επιμείνει ε, από κοινού να υπάρχουν δικαιώματα αποζημίωσης σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στις ε, διευρωπαϊκές διεθνείς μεταφορές. Ναι, να Πρόεδρε, ότι στην υπάρχουσα νομοθεσία υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να μην εφαρμόσουν τον κανονισμό για τις εθνικές μεταφορές με σιδηρόδρομο. Και πολλές χώρες, υπερβολικά πολλές κατά την άποψή μας, έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα αυτό. Είναι ένα από τα αισθήματα που θα μας απασχολήσουν. Ξέρετε ότι υπάρχει νομοθετικό κείμενο το οποίο σύντομα θα προχωρήσει. Θα αποτελέσει λοιπόν αντικείμενο και άλλων ακροάσεων αυτό ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χρειαζόμαστε, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία, έτσι. Διότι εμείς στη Γαλλία έχουμε τη μετάφραση του κυρίου Μακχό ε, για τα λεωφορεία, έτσι. Και δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα στο συγκεκριμένο τομέα. Ναι να βλέπουμε την κίνηση και και συγκεκριμένων επενδύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, πήγαμε πολύ γρήγορα σήμερα. Πήγε πολύ γρήγορα η ψηφοφορία. Οπότε ε, θα διακόψουμε ως τις 11 για να έχετε το χρόνο ε, να φωνάξετε και τους συναδέλφους να είναι εδώ στις 11 διότι έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές του ΔΕΔ. Ε, θα τα ξαναπούμε εδώ στις 11. Ευχαριστώ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε εκ νέου την ε, συνάντηση. Είμαστε στο σημείο 18. Ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές ε, των Ευρωπαίων Συντονιστών ε, των Ευρωπαϊκών Διαδρόμων. θα συζητήσουμε ένα οριζόντιο πολιτικό ζήτημα αφορά όλους τους διαδρόμους, πώς θα ενισχύσουμε τα συστήματα έξυπνων μεταφορών ε, απέναντι στην, ε, στο θέμα της εξάλληψης των ανθρακούχων εκπομπών. Θα μιλήσουμε για τον διάδρομο της Βαλτικής ε, και Αδριατικής. Ήταν να μιλήσουμε για αυτόν μάλλον, αλλά ο κύριος Μπόντε Βάιν δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Ζητή συγγνώμη γι' αυτό. Υπάρχει ο διάδρομος του Ατλαντικού που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Ζέκη. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κύριε Ζέκη. Και βεβαίως ο σκανδιναβικός και μεσογειακός διάδρομος με τον κύριο Κόξ. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Ε, αναμένουμε με ανυπομονησία την παρατήρηση την παρουσίασή σας. Έχετε 15 λεπτά ο καθένας, δηλαδή χρόνος υπάρχει ούτως ή άλλως σήμερα το πρωί. Θα μπορέσετε να παρουσιάσετε λοιπόν τις απόψεις σας. Στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση με τους ε, δύο εισηγητές, ο κύριος Ερτούγκ και ο κύριος Πίπερ που είναι οι μόνιμοι εισηγητές ε, για το ζήτημα αυτό. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε για άλλη μια φορά εδώ κάθε χρόνο, όποτε έχουμε τη δυνατότητα, κυρία, κυρία Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι να έρθουμε εδώ. Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το θέμα της λογοδοσίας, να λογοδοτούμε για αυτά που κάνουμε. Και το δεύτερο είναι το θέμα της κοινοβουλευτικής εποπτείας ε, και παρακολούθησης που είναι καθήκον δικό σας. Θα χωρίσω τα σχόλιά μου σε δύο σκέλη. Θα αναφερθώ, όπως είπατε και εσείς, ε, νομίζω σε μια διαφάνεια χωράνε όλα. Ε, θα αναφερθώ λοιπόν σε κάποια οριζόντια ζητήματα που αφορούν όλους τους ε, διαδρόμους. Ε, οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, άλλωστε εκπονήσει μια σειρά από κείμενα, issues paper, ε, για να καταλάβουμε καλύτερα το όλο ζήτημα. Και το δεύτερο σκέλος της παρουσίασης θα αφορά αποκλειστικά τον διάδρομο στο Σκανδιναβικό και της Μεσογείου. Ε, γενικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και της πρόκλησης αυτής. Ε, η COP21 στο Παρίσι και η Συμφωνία των Παρισίων ε, είναι πλέον για μας ο στόχος, έθεσε τους στόχους για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε και το Μάρτιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει έως το 2030 μείωση 40% των εκπομπών, δεσμευτικός στόχος. Και μεταφορές είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εκπομ... παράγοντας εκπομπών διοξείδου του άνθρακα και τα δύο τρίτα προέρχονται από τις οδικές μεταφορές, αλλά έχουμε αύξηση και στις αερομεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ε, Αντίθετα με τους άλλους τομείς, ε, δυστυχώς για τις μεταφορές έως το 2008 παρά την καινοτομία, τις καινοτομίες, τους νέους κανονισμούς, τους κανόνες για τα καύσιμα ε, ε, έχουμε τόσο πολλές μετακινήσεις, τόσο μεγάλη αύξηση των μετακινήσεων που τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι το 1990 αντίθετα με τους άλλους τομείς και με τους στόχους που έχουν τεθεί τώρα και τους περαιτέρω στόχους για το 2050, αυτό που είναι προφανές είναι ότι έχουμε τους φιλόδοξους αυτούς τους στόχους 2030, του 2040, 2050. Για να πετύχουμε το στόχο του 2050 όμως θα πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή της τάξης του 67% σε ό,τι αφορά τις εκπομπές στον τομέα των μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για πολιτικές αλλαγές ριζικές και όχι πλέον απλά διαχείριση. Ε, δεν θα σας πω τίποτα καινούριο βέβαια, αλλά είναι ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει ε, για την εξάλληψη των ανθρωπούχων εκπομπών. Χρειάζεται, χρειάζεται δημόσιες πολιτικές γι' αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στο modal shift, ε, να απομαχαινθούμε από τις, ε, ε, τα μέσα μεταφοράς τα οποία μολύνουν περισσότερο. Αυτή η μετάβαση λοιπόν πρέπει να λάβει χώρα να πάμε προς το σιδηρόδρομο, να πάμε προς τους, στις εσωτερικές πλωτές οδούς και από εκεί και πέρα το δεύτερο ζήτημα είναι η εναλλακτικά καύσιμα με ψηφικές ενέργειες, ηλεκτρικά οχήματα, υδρογόνο. Υπάρχουν πολλές μελέτες για τις εναλλακτικά καύσιμα και στο δικό μου διάδρομο ε, υπάρχουν κάποια πιλωτικά τεστ τα οποία λαμβάνουν χώρα. Τώρα, το, άλλο, το δεύτερο ζήτημα είναι πώς θα ε, κινητοποιήσουμε το EFSI και το Connecting Europe τα δάνεια, όπως περιπτώσει, ε, προέρχονται από αυτά τα ταμεία, δεν πρόκειται για ταμεία, και για δάνεια και όχι για ε, ενισχύσεις. Ε, Βεβαίω δεν αφορά αυστηρά τον τομέα των μεταφορών, αλλά στην οριζόντα του 2020 επίση υπάρχει ένα σκέλο που μα αφορά. Προσπαθούμε λοιπόν σε οριζόντιο επίπεδο να δούμε πώ θα μπορέσουμε να βρούμε του κατάλληλου μοχλού για να περάσουμε από μια αλλαγή σταδιακή που δεν έχει φέρει αποτέλεσμα ε, σε κάτι πιο φιλόδοξο, πιο ριζικό ε, για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Το δεύτερο οριζόντιο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ ε, είναι τα συστήματα έξυπνων μεταφορών. Είναι μια πολύ σημαντική τάση αυτή που έχει να κάνει την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση. Πρόκειται για σαφείς τάσεις οι οποίες θα ενισχυθούν στον τομέα των μεταφορών πρέπει να βγούμε λίγο από τα στεγανά. Ε, αν θέλουμε να δούμε ε, τις μεταφορές μέσα των, των έξυπνων αυτών συστημάτων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συγκλίνουμε και με συστήματα έξυπνης ενέργειας, ε, συστήματα νόσιμης ενέργειας και αυτό βεβαίως επικαλύπτεται και με τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ε, δίκτυα ψηφιακά, οπτικών ινών κτλ. Όλα αυτά πάνε μαζί ε, μέσω του χρήστη, μέσω του οχήματος, μέσω της υποδομής. Στο έγγραφο ITS λοιπόν, ε, για, τις, για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών δηλαδή, ε, επικεντρωθήκαμε στην σχέση μεταξύ οδηγού και οχήματος, οδηγού και χρήστη, ε, οχήματος και χρήστη. Από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα της επικοινωνία μεταξύ οχημάτων, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κυκλοφορία, την ασφάλεια στους δρόμους, η Ολλανδική Προεδρία έκανε κάποια σχετικά πειράματα πέρυσι. Πώ μπορούν αυτά τα συστήματα να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η τρίτη διάσταση είναι η επικοινωνία μεταξύ του οχήματο και τη υποδομή. Και το τρίτο είναι η διαχείριση των big data. Όλη αυτή, όλη αυτή η συνεχής ροή δεδομένων, επεξεργασία των δεδομένων αυτών που αποστέλουν στη συνέχεια στους διάφορους διαχειριστές συστημάτων και τους χρήστες των συστημάτων έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των υποδομών. Είναι εύκολο να τα λέει κανείς αυτά, αλλά δύσκολο να τα κάνει. Πιστεύουμε πάντως, είμαστε πεπισμένοι και το είδαμε στους διαδρόμους μας, ότι είμαστε ε, ένα πολύ καλό πεδίο πειραματισμού. Ε, υπάρχουν δυνατότητες αυτή τη στιγμή προσαρμοσμένες από τα υπάρχοντα δίκτυα ε, διασυνδέσεων που έχουμε σε οργανωτικό, σε πολιτικό επίπεδο, έτσι ώστε να γίνουν σωστές συζητήσεις ανάμεσα στους σωστούς ανθρώπους διασυνοριακά ε, ή διαπεριφερειακά. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ε, μία ε, προσέγγιση η οποία δεν έχει σύνορα. Είναι σημαντικό αυτό και για την κλιματική αλλαγή και για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών έχουμε ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούμε να καλέσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους εντός μίας δομής. Ε, όταν λοιπόν κάποιος έχει ε, μια καλή ιδέα ε, για την κλιματική αλλαγή, για τα έξυπνα συστήματα, θα πρέπει αυτό να τα εκμεταλλευτούμε, να το συνδυάσουμε. Συνέργειες είναι αυτό που χρειαζόμαστε, συνέργεια είναι αυτό που χρειαζόμαστε ε, θα ήθελα τώρα να περάσω στο θέμα του ε, διαδρόμου του Σκανδιναβικού και της Μεσογείου. Είναι το, ο άξονας βο, βορρά-νότου. Ξεκινάμε στα σύνορα ε, Ρωσίας-Φιλανδίας, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, ε, Βαλτική, Βόρεια λιμάνια ε, της Γερμανίας, Βερολίνο, Μόναχο, Αυστρία, Ιταλία, Σικελία, Μάλτα. Επτά κράτη-μέλη και η Νορβηγία συμμετέχουν 8 χώρε δηλαδή. Για να καταλάβετε λίγο πριν ως πρόκειται μιλάμε για 9.300 χιλιόμετρα σιδηρόδρομου στο δίκτυο αυτό, 6.300 χιλιόμετρα οδικών αξώνων, 19 αεροδρόμια, 25 λιμάνια και 44 σταθμοί ε, οδικών μεταφορών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Έχουν εγκριθεί, έχει εγκριθεί το δεύτερο σχέδιο δράσης, έχουν εγκριθεί από τις κυβερνήσεις αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη το έχουν εκπονήσει αυτό, αλλά και με τους ε, βασικούς ευλεκόμενους φορείς. Πρέπει, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα σημεία συμφόρησης, στάζουμε τα ζητήματα ε, προσθέμενης αξίας και εδώ επικεντρωνόμαστε στο ε, τούνελ του Μπρένερ από την ε, Ιταλία στην Αυστρία και τη Γερμανία όταν ολοκληρωθεί αυτό το τούνελ 64 χιλιόμετρα από την Φορτέντσα στο Ίνσμπρουκ από την Ιταλία στην Αυστρία λέει θα είναι το μεγαλύτερο τούνελ αυτού του είδου στην Ευρώπη και στον κόσμο. Βεβαίω νομίζω ότι οι Κινέζοι ετοιμάζουν κάτι ακόμα πιο φιλόδοξο στο άμεσο μέλλον. Αυτό ο διάδρομο είναι ήδη προχωρημένος. Ε, το τούνελ έχει προχωρήσει ήδη 16 χιλιόμετρα ε, γίνεται, υπάρχει ένα μέρος που είναι ε, βεβαίως ε, ε γίνεται, είναι ένα τούνελ ε, το οποίο είναι πειραματικό, είναι διερευνητικό 64 χιλιόμετρα λοιπόν προς το βορρά 64 χιλιόμετρα προς το νότο 64 χιλιόμετρα ε, διερευνητικό τούνελ στη μέση ε, για έρευνες συνολικά 220 χιλιόμετρα ε, να σας πω ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε υπογράψει όλες τις συμβάσεις για 80% του τούνελ. Ε, και αυτό έχει, ε, λαμβάνει χώρα λόγω της δέσμευσης της πολύ ισχυρής της Κομισιόν από το 2007 έχουμε διαθέσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ 40% των εξόδων ε, έχουν διατηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει επιστροφή πλέον και πάμε καλά από εκεί πέρα θα δούμε πώς ε, αυτό το τούνελ θα ολοκληρωθεί στην επιχειρησιακή φάση. Θα αργήσει ακόμα αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα σχέδιά μας. Θέλουμε να προωθήσουμε project τα, τα, για τα οποία είμαστε περήφανοι όταν θα, παρουσιάζουμε, όταν θα παρουσιάζουμε τα επόμενα χρόνια. το δεύτερο μεγάλο project αφορά τη Βαλτική. 19 χιλιόμετρα από τη Δανία στο Φέρμαν Island. Ε, θα δημιουργήσουμε εδώ μια περιοχή από το Αμβούργο ουσιαστικά, ε, την Κοπενχάγη, το Μάλμοε έως και στη Στοκχόλμη και ίσως και ως το Γκέτεμπορκ και, το, και μέχρι και το Όσλο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το project θεωρείται από όλους τους υπουργούς μεταφορών της περιοχής, ακόμα και αυτοί που δεν είναι Δανείοι ή Γερμανοί, θεωρούν ότι είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση όπου μπορούμε να προχωρήσουμε τις τελευταίες 12 μήνες ε, ε, δεν έχουν δοθεί ακόμα όλες οι άδειε. Ε, στη Γερμανία, στο Σλέσβι Χόλσταν υπάρχουν αντιδράσεις και πρέπει να σεβαστούμε τις αντιδράσεις και των πολιτών. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αψηφίσουμε, να μην σεβαστούμε τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει νωρί τη διαδικασία να το κάνουμε αυτό, να ξεκινήσει ο διάλογος με τους τοπικούς πληθυσμούς μπορεί να πάρει 5, 6, 7 χρόνια ε, να ξεπεράσουμε τα διοικητικά, τα νομικά ζητήματα, να ξεκινήσουμε όμως νωρίς για να μην συσσωρεθούν τα προβλήματα ε, για τέτοιου είδους μακροπρόθεσμα σχέδια. Το δεύτερο μεγάλο σχέδιό μας είναι ε, σιδηροδρομικό εντός της Γερμανίας. Δεν είναι διασυνοριακό αυτό, αλλά έχει επιπτώσεις και διασυνοριακά και επηρεάζει κυρίως τη Γερμανία. Όλες, όλα τα λιμάνια της Βαλτικής το Bremenhaven, το Αμβούργο, το Λούμπεκ, το Ρόστοκ ε, φέρνουν ε, αγαθά προϊόντα ε, στην ενδοχώρα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω σειροδρόμων. 48% γίνεται ήδη σιδηροδρομικά. Είναι το μεγαλύτερο στη Γερμανία. Όταν εξετάζουμε λοιπόν τις δυνατότητες που υπάρχουν, το πρόβλημα είναι ότι από την Ζηλανδία στην Χαν, στο Χανόβερ Υπάρχει ένα πρόβλημα δυνατοτήτων στο γερμανικό σύστημα. Βεβαίω είναι ένα γερμανικό πρόβλημα αυτό, αλλά μιλάμε για κάτι που έχει πτώσει σε όλο το δίκτυο. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε αυτό το γερμανικό θέμα, να το φέρουμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα, διότι οι επιπτώσει αφορούν το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο ζήτημα που εξετάζουμε, και θα τελειώσω με αυτά τα δύο ζητήματα, είναι συνοδευτικά μέτρα και διαδικασία προγραμματισμού. Σε ό,τι αφορά συνοδευτικά μέτρα, και εδώ αναφέρομαι σε ζητήματα όπω ε, τα διόδια, το πώς θα περάσουμε από τον οδικό στο σιδηροδρομικό, ε, στο δίκτυο. Ε, εξετάζουμε ε, το, την αρχή του ο χρήστης πληρώνει για το θέμα της συμφόρησης. συμφόρησης. Ε, βεβαίως μπορεί κάποιος να κάνει τα σχέδια, υπάρχει ο υδρολόγος, υπάρχει ο γεωλόγος, υπάρχουν οι χρηματοδότες, υπάρχουν οι προγραμματιστές. Όμως για να είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η πολιτική, διότι όλοι γνωρίζουμε, ο καθένας πιστεύει ότι αυτό που κάνει ο δικό του τρόπο είναι ο καλύτερο. Όταν γίνει μια σύνδεξη Αυστριακών, Ιταλών, Γερμανών, ο καθένα ε, λέει ε, ότι αυτό που έχει κάνει ω τώρα είναι το καλύτερο. Ε, θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν μια λογική κοινή για όλο τον διάδρομο, αλλά δεν είναι εύκολο. Όλοι έχουν συνεισφέρει. και φανταστείτε να επενδύσουμε δισεκατομμύρια λεφτά των φορολογουμένων για ένα υπέροχο project όπως ε, αυτό, αλλά τελικά να συνεχίσουμε να έχουμε δύο εκατομμύρια φορτηγά τα οποία να περνάνε από τον Μπρένεν και να μολύνουν αυτήν την υπέροχη περιοχή των Άλπαιων. Ε, αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Μέρος της διαδικασίας λοιπόν είναι να μοχλεύσουμε την αλλαγή μέσω άλλων εργαλείων. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να φυτέψουμε αυτό τον σπόρο. Δεν είναι δικό μα ούτε ο σπόρο ούτε το έδαφο, αλλά ε, έχουμε μια προοπτική. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι προφανέ. το ξέρουμε, το ξέρετε κι εσεί διότι είστε ε, εκλεγμένοι. Όταν εμφανίζεται ένα μεγάλο project, το οποίο έχει μια μακρά περίοδο κατασκευή, ε, έχει πολλέ επιπτώσει για τι τοπικέ κοινωνίε. πρέπει να ακουστούν οι τοπικέ κοινωνίε, Είναι σημαντικό πρέπει να ε, διαθέσουμε χρόνο ε, να μπορέσουμε να μετριάσουμε τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να βρεθεί ε, ένα, μια συνένεση. Και αυτό απαιτεί όλοι μας, αλλά κυρίως οι αρχές σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, όταν προσυπογράφουν ένα ευρωπαϊκό deal, να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση σε τοπικό επίπεδο νωρίς νωρί, πολύ νωρί, διότι ξέρουμε ότι παίρνει χρόνο. Και αν δεν ξεκινήσει κανεί νωρί, τελικά καταδικάζουμε αυτά τα project να είναι απλά ε, ένα μπάλωμα και όχι ένα δίκτυο, διότι δεν θα είναι ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένο το project παρά τι ε, πολύ σημαντικέ επενδύσει. Αυτά ήθελα να σα πω. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Euh, Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία και αισιόδοξη παρουσίασή σας. Ήταν όλα πολύ κατανοητά. Δίνω το λόγο στον κύριο Σέκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής μας και Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόσο για να υπάρξει μια ενημέρωση σχετικά με το τι συμβαίνει στο θέμα, των, ε, στο θέμα του Ατλαντικού Διαδρόμου και για να συζητήσουμε ορισμένα σημαντικά οριζόντια θέματα μαζί σας που σχετίζονται με την κοινοτομία όπως είπε και ο συνάδελφος Πατ Κόξ, με ειδική επικέντρωση στην ε, χρηματοδοτική καινοτομία. Εγώ θα κάνω την παρουσίασή μου λίγο ανάποδα από ότι ο κύριος Κόξ, Κόξ ο οποίος μας μίλησε για τον σκανδιναβικό μεσογειακό διάδρομο. Εγώ θα σας μιλήσω για τον Ατλαντικό που έχει μια ιδιαίτερη θαλάσσια διάσταση ε, καθώς συνδέεται με πολύ σημαντικά λιμάνια, συνδέεται με τον ε, ε, διάδρομο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών 4 και όταν ολοκληρωθεί, ο διάδρομος αυτός θα παίξει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στις επιβατικές μεταφορές, αλλά κυρίως στις εμπορευματικές. Έχει τέσσερις διασυνοριακές, ε, διασυνοριακά τμήματα, τέσσερις ε, διελεύσεις συνόρων και συνδέει όπως και οι βαλτικές χώρες έχει δύο ε, βασικούς, ε, βασικά σκέλη, το UIC και τον Ιβυρικό. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό η πορτογαλική και η ισπανική κυβέρνηση να έρθουν σε συμφωνία και να βρουν έναν τρόπο να επιλύσουν το, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και προκειμένου να υπάρξει ε, καλύτερη αποτελεσματική, αποτελεσματικότερη ε, ένταξη στον ευρωπαϊκό διάδρομο. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν και εν ώψη της νέας ε, χρηματοδοτικής περίοδου. Η κατάσταση στον ε, διάδρομο ε, αποτυπώνεται εδώ σε αυτή τη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ ποια κομμάτια έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, σε κυκλοφορία ποια πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα και ποια ε, πλήττονται από καθυστερήσεις. Και υπάρχει και το σημαντικό στοιχείο της έλλειψης διασύνδεσης Ισπανίας και Πορτογαλίας, το οποίο προσπαθούμε να υπερβούμε Παρ' όλα αυτά, όλε οι χώρε, τόσο τη Ιβηρική Χερσονήσου όσο και η Γαλλία, καταβάλουν σημαντικέ προσπάθειε. Ποια είναι τα βασικά επιτεύγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι η ταχεία γραμμή Tour Bordeaux έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, τον Ιούλιο θα τεθεί σε κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα ε, στον κόσμο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το LGTT, που είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αποδείχθηκε πως ήταν πολύ χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση. Το οποίο και θα χρηματοδοτήσει τις εμπορευματικές και τις τοπικές μεταφορές επίσης. Επίσης, άλλο επίτευγμα είναι η έναρξη λειτουργίας ενός Ταμείου για την προσβασιμότητα στους λιμένες στην Ισπανία, το οποίο υποστηρίχθηκε από το ΕΦΣΙ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση για την συγχώνευση, την χρηματοδοτική συγχώνευση διαφόρων έργων προκειμένου να επιτύχουμε αποτελεσματικότερη εφαρμογή και αξιοποίηση του ΕΦΣΥ. Το Ταμείο αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε, συστάθηκε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συγχωνευθούν κατά κάποιο τρόπο διάφορα μικρή, μικρά έργα σε ένα σύνολο έργων το οποίο διαχειρίζεται μία αρχή και ως προς τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΦΣΥ. Και τέλος, ένα ακόμη επίτευγμά μας ήταν το γεγονός ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση του έργου, ιδίως στην Ιβυρική Χερσόνησο, όπου υπάρχει μια διακυβερνητική ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας που ε, ασχολείται με θέματα διαλειτουργικότητας αλλά και η οποία ενημερώνει και ενημερώνεται συστηματικά και τακτικά όσον αφορά τους ε, κρίκους που λείπουν στον διάδρομο αυτόν. Χρηματοδοτικές επενδυτικές ανάγκες ανέρχονται σε 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές έχουν ήδη επενδυθεί 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρία από αυτά τα δισεκατομμύρια έχουν δοθεί από το ΣΕΦ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. αλλά και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία ε, βοήθησαν στο να εξευρεθούν επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων και να σημειώσω επίσης ότι ένα ποσό 7-8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρη συνδρομική διαλειτουργικότητα στην Ιβυρική ε, Χερσόνησο λόγω της διαφοράς του εύρους τροχών ε, στην ε, Ιβυρική Χερσόνησο και, την, ε, και το UIC. Αυτό το θέμα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής και ελπίζουμε να, να καταφέρουμε να το επιλύσουμε. Να περάσω τώρα στο επόμενο τμήμα της παρουσίασής μου, το οποίο αφορά την καινοτομία ε, ως προς τη χρηματοδότηση. Όλα αυτά βεβαίως πηγάζουν από τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες που υπάρχουν προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους και τις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Ε, εκτιμάται ότι οι επενδυτικές χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται σε ύψος 750 δισεκατομμύρια ευρώ που βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλυφθούν από τα διαθέσιμα ταμεία. Άρα λοιπόν χρειάζεται να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια, γνωρίζετε ότι αυτό είναι πάντοτε πλέον ένα από τα συστατικά στοιχεία, και να δοθούν όχι απαραίτητα κίνητρα για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, αλλά να βελτιωθεί το πλαίσιο εντός των οποίων αυτές μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτός ήταν και ο στόχος της έκθεσης CBS, η οποία ολοκληρώθηκε, εκπονήθηκε πριν από ορισμένα χρόνια, που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο και σε εσά, επί της οποίας εργαζόμαστε ακόμη όχι μόνο για να παρακολουθούμε τι εφαρμόζεται, αλλά για να μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα για τα προβλήματα που ανακύπτουν. Γνωρίζετε ότι τέσσερα ήταν τα πεδία που μας ενδιέφεραν κυρίως, στα οποία επικεντρώσαμε την προσοχή μας. Πρώτον, ενίσχυση της, ε, του σχεδιασμού των, των έργων, ε, οικοδόμηση ικανοτήτων, συμβουλευτικό κέντρο, αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας στις δημόσιες προμήθειες, στις ε, κρατικές επιχορηγήσεις, διεύρυνση της χρηματοδότησης ε, μέσω της χρήσης διαφόρων πηγών και ε, θετικά αποτελέσματα, ένα θετικό περιβάλλον όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τη διαχείριση των ε, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα και την εμπλοκή των ε, ενδιαφερομένων πλευρών. Αυτά λοιπόν ως προς το CBS. Να σας πω τώρα ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την δημοσίευση της έκθεσης CBS και έπειτα. Όσον αφορά την υποστήριξη του σχεδιασμού των ε, μεταφορικών έργων, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε καλύτερα project που θα ε, ε, εμπλέκουν περισσότερο και τους ιδιώτες επενδυτές σε αντίθεση με ό,τι γινόταν παλαιότερα που τα θέματα αυτά ήταν αρμοδιότητας και ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για τις κρατικές αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ε, ΣΔΙΤ αλλά και για τη νέα ε, προσέγγιση ε, που είναι γνωστή ως συγχώνευση χρηματοδοτικών πηγών που ορίζει η νέα προσέγγιση ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της τεχνικής και της χρηματοδοτικής διαδικασίας που ακολουθείται για κάθε έργο. Όλα αυτά βεβαίως ε, υποστηρίζονται από το Τζάσπες, από, την, από το κέντρο ε, παροχής συμβουλών κτλ. κτλ. Δεύτερο, ε, δεύτερο στόχος ήταν να αντιμετωπιστούν βασικά διοικητικά ζητήματα. Υπήρξε η πρωτοβουλία για την ενιαία θηρίδα, η οποία συστήνεται και δημιουργείται όπου μας δόθηκε βεβαίως η δυνατότητα. Ε, αναθεώρηση των κανόνων κρατικών επιχορηγήσεων και ε, fast track ε, εκτέλεση των έργων του ΕΦΣΥ και αναθεώρηση και χαρτογράφηση της διαδικασίας αδειοδότησης θέμα για το οποίο εκπονήθηκε πολύ πρόσφατα και μια μελέτη η οποία και θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες και στην οποία ε, περιλαμβάνονται και ορισμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσαν να επιληθούν ορισμένα προβλήματα που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ε, ιδίως στις διασυνορικές περιοχές. Ε, για τις, για τις γλώσσες, για, τα, την σήμανση κτλ. κτλ. Διεύρυνση χρηματοδότησης και ναι, της χρηματοδότησης. Στόχος μας είναι να κινηθούμε σε μια πιο, και... μια πιο καινοτόμα προσέγγιση, το blending, δηλαδή η προσπάθεια να συγχωνευτούν διάφοροι πόροι προκειμένου να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος. Πρόκειται μάλιστα, ο, ο Ατλαντικός διάδρομος είναι ο πρώτος ο οποίος χρηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο. Μιλούμε για δάνεια ε, της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μιλάμε για κονδύλια ε, του ΕΦΣΙ, ε, μιλούμε για ιδιωτικά κεφάλαια. Όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η χρηματοδότηση του έργου. Και στο τέλος αυτής της διαδικασίας, της συγχώνευσης και του συνδυασμού, δίνεται και υπογράφεται και η συμφωνία μεταξύ των εταίρων. Και με αυτό επανέρχομαι και στο ζήτημα της ε, ποιότητας των έργων. Γιατί αν χρειάζεται να ε, πείσει κανείς μια εμπορική ή επενδυτική τράπεζα, χρειάζεται βεβαίως να έχει καταρτιστεί ένα άρτιο έργο από τεχνικής άποψης και αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να εξετάσουμε τα μεγάλα έργα υπό μια διαφορετική σκοπιά. Ε, αναφέρομαι στη δυνατότητα κατάτμισης ενός πολύ μεγάλου έργου ε, όσον αφορά τις πλατφόρμες ε, επιμελητίας, για παράδειγμα, μπορούν τέτοιου είδους έργα να ενταχθούν στο ΕΦΣΥ. Και τέλος, επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, να πω κάτι για τον τρόπο ε, που λειτουργεί η χρηματοπιστωτική αγορά. Υπήρξαν κάποιες σοβαρές τροποποιήσεις ε, στον κανονισμό για την φερικιότητα 2 και έχουμε ήδη περιπτώσεις μακροπρόθεσμων ε, στρατηγικών επενδυτών οι οποίοι έχουν εκφράσει την, ε, το ενδιαφέρον τους για το έργο μας ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση του κανονισμού Βασιλεία 3 που θα διευκολύνει την μόχλευση και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων ε, Βεβαίω υπάρχουν πολλά πράγματα που χρειάζεται να γίνουν έως τον, ε, το φθινόπωρο. Μιλώ εκ μέρους και του κυρίου, κυρίου Μπόντεβικ που δυστυχώς δεν μπόρεσε σήμερα να είναι μαζί μας για λόγους υγείας. Παρ' όλα αυτά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς εσάς για τη βοήθεια που μας παρέχετε ε, καθώς προσπαθούμε στο έργο μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τις δύο αυτές παρουσιάσεις που ήταν πολύ σαφείς και που περιλαμβάνουν και περιγράφουν πολλές προκλήσεις. Και όλο ένα τίθεται το ζήτημα των επενδύσεων αλλά θα επανέλθουμε αργότερα στο ζήτημα αυτό. Ας ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση, δίνοντας το λόγο στον κύριο Βιν Βαντεκάμπ. Ε, μάλλον στον εισηγητή πρώτα απ' όλα, Ισμαήλ Ερτούγκ. Okay, ε, καλά είναι μέχρι στιγμή τα πράγματα. Ευχαριστώ και τους δύο παρουσιαστές, κύριε Κόψ και Σέκη. Πρέπει να επαναλάβω ότι αυτές οι 20 κατευθυντήριες γραμμές και αυτή η δομή των διαδρόμων και οι κατευθυντήρες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, είναι η καλύτερη ιδέα που είχαμε τα τελευταία χρόνια ε, τη βρίσκω πολύ καλή και ο συζητητή και ο συντονιστής και έχω την εντύπωση ότι όταν δεν υπάρχουν προβλήματα κανείς δεν ε, φωνασκεί. Οπότε νομίζω ότι κάνετε τη δουλειά που κάνετε με τους υπουργού και τους ομολόγους σας ε, στην, ε, στα κράτη και όταν τα πράγματα γίνονται έτσι είμαστε και εμείς ικανοποιημένοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά από την εμπειρία σας θα ήθελα να μάθω το εξής. Πριν 4-5 χρόνια είχαμε συζητήσει αυτό το νομοθέτημα και τότε είχαμε δυσκολευτεί να περάσουμε την ιδέα αυτή από το Συμβούλιο. Τις πλατφόρμες, ε, τις ε, διαδρομές ε, πλατφορμών και στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει μια δυσκολία να πείσουμε τους ομολόγους μας στο εθνικό επίπεδο να έρθουν, να συζητήσουν. Και εσείς τώρα πώς θα περιγραφείτε, τι εμπειρία έχετε. Νομίζω τώρα έχουν συμφωνήσει. Ε, τυχόνευσαν την ιδέα ε, την ευρωπαϊκή αυτή. Έχω δίκιο, έχω άδικο, αυτή, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση για όλο τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Ισμαήλ Ερτούγκ. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Βίμ Βαντεκάμπα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε και ο κύριος Έρτογκ. Ε, ε, είναι ε, εξαιρετική η παρουσία σας σήμερα εδώ και μας δώσετε μια πολύ καλή εικόνα των πραγμάτων με τον οποίο έχουμε να ασχοληθούμε εδώ και είναι πολύ καλό πιστεύω που έχει εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε και άλλους συντονιστές εδώ και Πιστεύω ότι η εικόνα είναι πολύ καλή. Διότι πρέπει κανείς να βγει από τους δικούς του διαδρόμους και να δει την ευρύτερη εικόνα, τη γενικότερη εικόνα. Και χαίρομαι που βλέπω τον Πατ Κόξ εδώ ε, και που έχει αυτή την προσέγγιση να εξετάσει τα νέα στοιχεία πολιτικής, την απαλλαγή από τις ανθρακούς εκπομπές, τα ΕΦΗ, συστήματα μεταφορών ε, και που μελετά την ένταξη αυτών στα ε, προγράμματα διευρωπαϊκών δικτύων, διότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε τεράστιες γενικές διευθύνσεις που εργάζονται ε, σε μόνες τους ουσιαστικά μέσα σε μια φούσκα και μου αρέσει που έχετε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα ζητήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε φυσικά. Πριν από μερικούς μήνες συζητήσαμε μια έκθεση του Ελεκτικού συνεδρίου για τις ε, επενδύσεις ε, στις θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια στην Ευρώπη. Ήταν ε, κρίσιμη σημασία η έκθεση αυτή. Εξέταζε διάφορα ισπανικά λιμάνια, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του κ. Σέκη. Δηλαδή, έχουμε ένα μοντέλο, έχουμε μια γραμμή, όπως είπε και ο Ισμαήλ, και δεν λέω να παρεκκλίνουμε από αυτήν, όχι, να μείνουμε σε αυτήν, αλλά οι επενδύσεις επίσης θα πρέπει να έχουν κάποια νομιμοποίηση. Θα πρέπει δηλαδή ε, θα πρέπει να κάνουμε κάπως ε, τα πράγματα ώστε να περνάνε τα εμπορεύματα από τα λιμάνια. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Πριν δύο χρόνια συζητήσαμε εδώ μια έκθεση για μακροεπενδύσεις ε, στις αστικές διασυνδέσεις που επίσης δημιούργησε διάφορες αμφιβολίες, διάφοροι δήμοι και δημοτικά συμβούλια θέλαν τις δικές τους γραμμές ε, μετρό χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν επιβάτες ε, για αυτές τις γραμμές. Ε, και αυτό με φέρνει στο θέμα των προτεραιοτήτων. Στην έκθεση του κυρίου Κόξ αναφέρεται ότι η Φιλανδία φαίνεται σαν να είναι στην άκρη του κόσμου ή στην άκρη της Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα στο Μάνχαεμ χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις ώστε να συνεχίσει η πόλη να είναι ε, ε, βιώσιμη. Ε, τι κάνει δηλαδή κανείς πάει στο Μανχάιμ και βλέπει τι μπορεί να κάνει για να κάνει τους κατοίκους πιο ευχαριστημένους ή πάει στη Φιλανδία δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Και μετά, όσον αφορά τις άδειες ε, ε, οικοδόμησης, ε, στην εισαγωγή του ο Πατκόξ αναφέρθηκε σε άδειε κτηρίων, ξανά και ξανά και πώς μπορούμε να βρούμε κίνητρα ε, και είπε ο κύριος Σέκη ότι θέλουμε ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης. Αλλά έχουμε και το εννέα. Το εννέα τι κάνει. Το εννέα, συγγνώμη. Ε, όπως κατάλαβα, ναι, το, το, το, το ε, ενιαίο σημείο εξυπηρέτηση στην Κομισιόν θα ήταν το εννέα. Το 9. Τελευταία ερώτηση. Ε, ο κύριος Κράμερο, Ισμαήλ και εγώ επίσης, επισκεφθήκαμε τη σύραγγα Μπρένα και ακούσαμε ότι η διάτρηση πάει μια χαρά, αλλά ότι οι οδοί πρόσβαση δεν πήγαιναν καλά. Είδαμε στο σύραγγα του Γοτάρδου, ε, τα, οι ε, οδοί πρόσβαση ήταν πολύ περίεργα φτιαγμένε. Δυστυχώ δεν μπορώ να περιμένω για την απάντηση, διότι το προσωπικό του ΕΛΚ και το δικό μου προσωπικό όμω θα είναι εδώ και θα ακούσουν την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βαντεκάμπα, κύριε Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ολλανδικά ακούσαμε, τώρα θα ακούσουμε γερμανικά. Καταρχά. όχι, τα Ολλανδικά μου δυστυχώ δεν είναι τόσο καλά. Τα Γερμανικά μου είναι καλύτερα. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω λοιπόν ε, του δύο συντονιστέ για την έκθεση. Είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον να μα ενημερώνετε για το τι γίνεται με του διαδρόμου. Και όπως είπε και ο, ε, ο Ισμαήλ Ερτούγκ, ε, είναι πραγματικά πάντο ε, πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε αυτούς τους χάρτες με τους σταθμούς των πόλεων, και την, των, των πόλεων που συνδέονται και τη χρηματοδότηση που απαιτείται. Ένα ερώτημα για τον κύριο Σέκη. Είπατε 750 δισεκατομμύρια. Είναι το συνολικό ποσό, έτσι, όχι μόνο το δικό σας ε, διάδρομο, αλλά για όλους τους διαδρόμους. Ωραία, εντάξει. Δεύτερον, είχατε εκδώσει κάποιες ε, συστάσεις για το πώς μπορούν να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια. Στο Connecting Europe Facility είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε ομόλογα έργου είναι πολύ δύσκολο όμως τελικά να ε, τα αποκτήσει κανείς αυτά ε, ή εν να, τα, να συσταθούν τέτοια ομόλογα. Υπάρχουν ωστόσο παραδείγματα όπου κάτι τέτοιο να στέφθηκε με επιτυχία. Και έχω και ορισμένα ερωτήματα για τον Πατ Κόξ. Πρώτον, για το ζήτημα των εκπομπών. Ε, πάντοτε μιλούμε για μια μετατόπιση των ροών ε, μεταφορών στις εσωτερικές πλωτές ή στις ισοδρομικές. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Ε, ιδίως οι εμπορευματικές μεταφορές μειώνονται, ε, οι εμπορευματικές ειδοδρομικές μεταφορές, γιατί λείπουν τόσο οι κόμβοι όσο πολλές φορές και η τεχνολογία για τη μεταφορά εμπορευμάτων από φορτηγά οχήματα σε σειρμούς τρένων. Έχετε κι εσείς αυτή την ε, εντύπωση. Επίσης, υπάρχει ένα δίκτυο για την ανάπτυξη ε, της διάδοσης των ε, ανανεώσιμων εναλλακτικών πηγών ε, ενέργειας. Τι συμβαίνει με αυτό. Και ένα ερώτημα για τον διάδρομό σας. Ε, για, για, και για τους δύο διαδρόμους εδώ που τα λέμε. Ε, ο Ατλαντικός διάδρομος αλλά και ο Σκανδιναβικό-Μεσογειακός ε, περιλαμβάνουν πολλούς λιμένες. Πιστεύετε ότι τα λιμάνια αυτά είναι επαρκώς εξοπλισμένα με υποδομές επεξεργασίας λιμάτων. Γιατί ε, έχει ακουστεί ότι πολλά λιμάνια στην Ευρώπη δεν έχουν τέτοιες κατάλληλες υποδομές και βεβαίως ε, φαντάζομαι ότι θέλουμε να αποφύγουμε την ε, περιττή ρήπανση μόλις του περιβάλλοντος. Και τελευταίο ερώτημα. ΑΕ που συνδέει βρέμι με ανόβερο. Πήρε πάρα πολλές αναβολές αυτό το έργο. Υπάρχει όμως πλέον κάποιο χρονοδιάγραμμα το οποίο να έχει τεθεί σε συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ, ο κύριος Κράμερ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις. Θέλω ιδίως να ευχαριστήσω τον Πατ Κόξ που μας παρουσίασε ολόκληρη την ε, διάσταση του θέματος. Οι μεταφορές είναι ο μοναδικός κλάδος στον οποίο οι εκπομπές αυξήθηκαν 28% από το 1990, ενώ η βιομηχανία μείωσε τις εκπομπές κατά 38% στο ίδιο διάστημα. Άρα είναι απόλυτη επιτακτική η ανάγκη ε, μετατόπισης των ε, ροών μεταφορών. Έχουμε και εμπειρία με, τον, με το τούνελ που θεωρώ ότι ήταν μια καταστροφή για την Ευρώπη και το περιβάλλον. Τέσσερις ε, χώρες υπέγραψαν την ε, συμφωνία του Λουγκάνο και εξ αυτών μόνο η Ελβετία ε, ακολούθησε και τήρησε τις δεσμεύσεις της. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί δεν κάνουν τίποτα εδώ και 20 χρόνια γιατί δεν υπάρχουν ούτε καν οι, ε, δεν υπάρχουν καν οι, τεχνολογίες. Στην Ιταλία ε, γίνεται απλώς ένα έργο διασύνδεσης, το οποίο όμως χρηματοδοτείται από την Ελβετία. Η Ιταλία δεν κάνει τίποτα και όταν πας εκεί ε, οι αρχές ε, σου δίνουν την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρονται καν. Παρότι έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτές τις συμφωνίες. στη Γερμανία, ρωτήσαμε τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος ομολόγησε ότι δεν υπάρχει ούτε καν η χάραξη ε, του, του, του αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει ε, το δικό δίκτυο με το Brenner. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά, το Ρήνο, Ιταλία. Και εγώ έχω θέσει το ερώτημα τι κάνετε για να παρακινήσετε τις ε, χώρες να ολοκληρώσουν πρώτα και κύρια αυτόν τον σημαντικότερο ε, ε, ε άξονα διάδρομο και μετά μπορεί να συζητήσουμε και για άλλα έργα στην Ιταλία ή στη Γερμανία τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν είναι ικανές οι χώρες αυτές να ολοκληρώσουν αυτό το βασικό έργο που έχει υπογραφεί και συμφωνηθεί πριν από 20 χρόνια. Είναι αποφασιστική σημασία. Για τον για το έργο Μπελκέρο. η γερμανική κυβέρνηση είχε πει εντάξει, άμα θέλουν οι Δανείοι το χρηματοδοτήσουν και το κατασκευάσουν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα διότι η ολόκληρη κυκλοφορία ε, περνάει μέσα από το Αμβούργο. Υπάρχει όμως και η άλλη σύνδεση μέσω του Ρόστοκ. Ρόστοκ, Γκέτσα, Νίκιόπινγκ. Είχαμε μάλιστα ε, αποφασίσει εδώ στο Κοινοβούλιο ε, να εξασφαλιστούν χρήματα για τον εξυγχρονισμό εκείνης της, ε, εκείνου του, διαδρόμου αλλά και εκεί εμφανίστηκαν οι Δανείοι με δικά τους προβλήματα και δικές τους αντιρρήσεις. Και τελικά καταλήξαμε στο να χρηματοδοτούνται έργα και για τις οδικές μεταφορές και για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Κάτι που βεβαίως δεν θα μας βοηθήσει στη μεταπιτώπιση των ροών μεταφορών. Για τα χρηματοδοτικά μέσα, ERS, EATMS και όλα αυτά Υπάρχουν προβλήματα ε, μη συμβατότητας το, το, του εύρου τροχών μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα των ε, των σειρμών να περνούν από, το ένα, από τη μία χώρα στην άλλη. Ή θα έχουμε πάλι το ίδιο παιχνιδάκι που θα λένε αρχές ότι όχι, δεν γίνεται να, να μπείτε στη δική μου χώρα γιατί δεν... Ε, ε, δεν είναι συμβατά, συμβατό το εύρος τροχών σας. Μπορείτε να μας ε, ε, πείτε ορισμένες περισσότερες πληροφορίες για το τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο. Ευχαριστώ κυρία Κλούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόσκη, τον κύριο Σέκη για τις συνεισφορές τους Εγώ ενδιαφέρομαι βεβαίω ε, για την Βόρεια Θάλασσα, Μεσόγειο, αυτό το, το, ε, το διάδρομο δεν είναι εδώ ε, σήμερα ο εκπρόσωπο για να το συζητήσουμε, αλλά εν πάση για τη χρηματοδότηση που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ε, ο κ. Σέκη αναφέρθηκε ε, στη συγκέντρωση για τη μόχλευση, είναι σημαντικό αυτό για τα μικρά project, μάλλον και τη μόχλευση για το pooling, μπορούν να συγκεντρώνονται ε, κάποια χρήματα, ε, να υπάρχει μια δεξαμενή, εν περιπτώσει, που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση πιο μικρών project. Και για την ενιαία θηρίδα και αυτό είναι μια πολύ θετική προσέγγιση. Να πω αυτή εξ αρχή ότι εγώ θεωρώ είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διάδρομη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ε, Βόρεια Φιλανδία, αλλά και άλλες περιοχές, η Ιρλανδία από που προέρχομαι, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η διασύνδεση με, το, με την καρδιά της Ευρώπης. Είναι σημαντικό και θετικό το ότι υποστηρίζουμε αυτούς τους διαδρόμους και το ότι προχωρούν τα διάφορα project. Ένα θέμα οριζόντιο, οι θαλάσσιες λεωφόροι, θαλάσσιες λεωφόροι δεν έγινε αναφορά σχετικά, υπήρχε μια ανησυχία ότι ενδεχομένως δεν θα υπήρχε ε, έτσι διασύνδεση μεταξύ των TNT και των λεωφόρων των θαλάσσιων. Ε, θα ήταν λογικό όμως να υπάρχει διασύνδεση. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Μπορείτε να σχολιάσετε από αυτού. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για τις εισφορές σας και αναμένουμε το φθινόπωρο την έκθεσή σας. Ευχαριστούμε κυρία Κλέον. Κυρία Μοντέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, δύο παρουσιάσεις αυτές. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ακούσαμε την Ολλανδία, τη Γερμανία και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Ατλαντικό. Ας πάμε λοιπόν στην Πορτογαλία. Εγώ είδα όλα αυτά που παρουσιάσατε και φυσικά διάβασα τα έγγραφα και έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι η διάσταση των θαλάσσιων μεταφορών όσον αφορά τις θαλάσσιες οδούς, τις λιμενικές υποδομές, την αποτελεσματικότητά τους τα συστήματα e-maritime όπως τα ονομάζουμε, τα καύσιμα ε, εναλλακτικής φύσης, ε, ε, το LNG. Πιστεύω ότι δεν έχετε εμβαθύνει επαρκώς σε όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν κάποια κενά όσον αφορά τη δημιουργία ναυτικών αντιπροσωπών. Πιστεύω ότι χρειάζονται νέα ε, προγράμματα ώστε ε, να ε, ε, δώσουμε περισσότερη σημασία στις προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, στο εμπόριο, στις αντιπροσωπείες των θαλασσιών μεταφορών, να επιμείνουμε για την, νομοθεσία, την περιβαλλοντική νομοθεσία για τα μεγάλα πλοία. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Ήθελα επίσης να επανέλθω, να σχολιάσω κάποια σημεία η αποθήκευση και η διανομή ε, LNG υγροποιημένου φυσικού ή αερίου Πιστεύω ότι οι χώρες που βρίσκονται προς το Ατλαντικό έχουν ένα δυναμικό το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα στο έγγραφα. Όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για τα εναλλακτικά καύσιμα, ε, πώς συνδέονται τα σχέδια αυτά και τα εθνικά σχέδια σχετικά με τα λεπτομερή εθνικά σχέδια για τις ε, θαλάσσιες οδούς. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό. Μετά, η αυτόνομη ε, περιφέρεια της Μαδέρας ε, και το λιμάνι της Μαδέρας που έχουν ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο ε, δεν γίνεται καμία αναφορά στο πρόγραμμα αυτό. Πιστεύω ότι η νησιωτική ε, διάσταση του Ατλαντικού δεν λαμβάνεται επαρκώς. Μπορείτε να μου απαντήσετε γι' αυτό. Ε, συγγνώμη τώρα θα κάνω περισσότερο ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Σέκη για το κομμάτι του Ατλαντικού. Στη συνέχεια τώρα Αναφέρουμε συχνά ε, κάποιες συνδέσεις, αλλά αναρωτιέμαι τι λείπει. Το πρόγραμμα ε, προοδεύει όπως έχει προβλεφθεί και έχει λάβει τις διαστάσεις που είχαμε προβλέψει. Εσείς τι πιστεύετε, είναι κρίσιμο το σημείο αυτό. Ε, μια άλλη παρατήρηση Ε, μια άλλη ερώτηση για τη βόρεια περιοχή της ε, Πορτογαλίας, εκεί που συνδέεται με τη Γαλλικία, δεν εντάσσεται στο διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά αυτό θα ήταν σημαντικό. Εσείς ε, τι λέτε για το γεγονό ότι δεν έχει συμπεριληφθεί. Δεν έχουν συμπεριληφθεί αυτές οι δύο περιοχές. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Merci beaucoup. Monsieur euh, Milterberg, c'était Merci. Ευχαριστώ Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή δουλειά που κάνατε ε, για τον διάδρομο αλλά και για τα issue papers η γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΜΚΟ για τη δράση ε, της, Κομ, της Κομισιόν ε, για το CITS είναι κάτι που με απασχολεί έχω ασχοληθεί με αυτό. Θέλω να σα ευχαριστήσω και για Πατκόφ για αυτό που έχετε κάνει για το ITS, για τα έξυπνα συστήματα ε, μεταφορών. Ένα πράγμα είναι σαφέ εδώ. Αυτό το έγγραφο συστήνεται ο ε, ε διάδρομος ITS να επεκταθεί και να καλύπτει όλους τους διαδρόμους. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συντονισμός. Θα πρέπει αυτή την πρόκληση να την ε, ε, αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη και ευρύτερη χρήση του ITS. Εφόσον λοιπόν πιστεύετε πρέπει να καλυφθούν όλοι οι ε, διάδρομοι, πιστεύετε πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός συντονιστής ευρωπαϊκός για το ε, ITS όπως έχουμε και το EMTS ή για τους τηλεοφόρους της θαλάσσης ε, επειδή στο έγγραφό σας αναφέρεστε στους, στα πειράματα, στα πεδία πειραμάτων και υπάρχει ήδη χρηματοδότηση από το ΣΕΦ για ένα σχετικό πρόγραμμα. Ποια είναι η άποψή σας για τις ανάγκες επενδύσεων. Μπορείτε να κάνετε μια αξιολόγηση πώ θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε παραδείγματο χάρη τα διασυνοριακά, τα ζητήματα που συνδέονται και με τι υποδομέ δεδομένων. Μπορείτε επίση να μα πείτε κάτι και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Ε, είναι σημαντικό που έχουμε αυτή την ενημέρωση εκ μέρους σας. Ακούσαμε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για τις, ε, τα έξυπνα συστήματα μεταφορών, για τη χρηματοδότηση, για την εξάλληψη των ανθρακούχων εκπομπών, αλλά δεν τελειώνει ένας διάδρομος εκεί που πιστεύουμε ότι τελειώνει. Εγώ είμαι από τη Βόρεια Σουηδία, στον χάρτη φαίνεται ο διάδρομος να σταματάει σε κάποια μεγάλη πόλη, Στοκχόλμη, Ελσίνκη, Όσλο. Όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ζωή και πιο βόρεια. Εάν δείτε το χάρτη, ε, θα δείτε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πλεονέκτημα με τους διαδρόμους αυτούς είναι ότι μπορούμε να δούμε το σύνολο της διαδρομής και βλέπουμε πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Όταν όμως δεν το βλέπουμε αυτό με ακρίβεια στον χάρτη, αν δεν φαίνονται όλες τις διασυνδέσεις, ο Παρκόκος το ξέρει, έχει πάει στη Βόρεια Σουηδία, αλλά οι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. 90% όλων των πρώτων υλών ε, προέρχονται από τη Βόρεια Σουηδία. Ε, υπάρχουν συμφορήσεις εκεί, σημεία συμφόρησης βόρεια από τις, της έξω από τους διαδρόμους που βλέπετε στο χάρτη. Πρέπει να προσθεθεί λοιπόν αυτός ο διάδρομος στο χάρτη. Ε, βεβαίως γίνονται κάποια πράγματα πειραματικά με τους διαδρόμους αυτούς. Ε, ο πράσινο, πράσινος κινητόδρομος ε, προς το Τρότχαιμ, όπου ε, έχει γίνει μια επένδυση για να υπάρχουν σημεία που να μπορεί κάποιο να φορτώσει με ηλεκτρική ενέργεια το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά όλα αυτά δεν αναφέρονται στο χάρτη. Γιατί το λέω αυτό, το λέω για παιδαγωγικού λόγου. Ε, εάν στη Βόρεια Σουηδία θέλω να εξηγήσω, θέλω να περασπιστώ μια επένδυση, ε, πρέπει να το δουν οι άνθρωποι πώ συνδέεται αυτό με του διαδρόμου. Από παιδαγωγική πλευρά, λοιπόν, σα το λέω, για να έχετε μεγαλύτερη υποστήριξη, να είστε πιο ακριβεί στου χάρτε. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσεν. Κύριε Ρικέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσει τους. Λοιπόν, το πρώτο που έχω να πω ήταν ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και ε, πρωτότυπες γιατί αποδεικνύουν ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη εικόνα των διευρωπαϊκών δικτύων. Συνήθως έχουμε την αίσθηση ότι όταν έρχονται οι συντονιστές των δικτύων μας παρουσιάζουν ε, ένα παιχνίδι με τουβλάκια ε, όπου κερδίζει αυτός που παίρνει τους περισσότερους πόντους και ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι ενώ εδώ είδαμε μια θεματική εικόνα των δικτύων τόσο στην οριζόντια διάστασή τους ε, από τον Πατκόξ όσο και για τον οικονομικό έλεγχο και τα ουσιώδη στοιχεία. Λοιπόν, η πρώτη παρουσίαση μας έδειξε ουσιαστικά ότι τα δίκτυα δεν είναι απλά ένα γεωγραφικό παιχνίδι και είναι σφάλμα να παρουσιάζονται έτσι. Η δεύτερη παρατήρηση που είχα να κάνω είναι ότι η αξία ενός ολόκληρου διαδρόμου είναι ανώτερη από, το επιμέρους, από αυτή, το αθροίσματος των επιμέρους μερών του. Διότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι με τα λέγκο, το παιχνίδι που, χτίζουμε σπιτάκια, ε, έχει ως αποτέλεσμα ε, κάτι πολύ ομορφότερο από ό,τι τα κομμάτια του, τα επιμέρους κομμάτια. Μόνο που δεν μπορούμε το κάθε κομμάτι να το διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Εξακολουθεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό τμήμα παρότι αποτελεί ένα κομμάτι συνόλου. Και όπως βλέπετε ε, το κάθε κράτος μέλος λέει και αυτό που αφορά το, το, τον εαυτό του, αλλά δεν δημιουργήθηκε αυτό για, αυτό. Ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε σε αυτή, σε αυτή, σε αυτή την ιδέα του οράματος Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι μπορούμε να, έχουμε, να επιτύχουμε κάποια συνοχή όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο, την οικονομική διαχείριση. Υπάρχουν επιχορηγήσεις, υπάρχουν ε, χρηματοδοτήσεις και μετά υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας. Υπάρχουν πολλά κομμάτια. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι δυνατή η συνοχή σε οικονομικό επίπεδο. Και μου φέρει και ενδιαφέρουσα η πρόταση που άκουσα ότι ουσιαστικά μπορούμε να αντιστρέψουμε τη γενική διαδικασία ε, όχι να λέμε δηλαδή πόσες επιχορηγήσεις υπάρχουν και θα σας πω τον προπολογισμό αλλά να βρίσκουμε τα χρήματα ας πούμε μέσω χρηματοδοτήσεων ε, ε, τραπεζικών ή ιδιωτικών ε, λοιπόν επενδύσεων και μετά να προσαρμόζουμε την επιχορήγηση. Το δεύτερο μου ερώτημα, ε, οι συντονιστές μας πιστεύουν ότι είναι ευκολότερο να υπάρχει γεωγραφική διαχείριση από τη θεματική. Γιατί έχω την εντύπωση ότι για πολιτικούς λόγους και λόγους διαφορών συμφερόντων η διαχείριση αυτή είναι γεωγραφική περισσότερο. Και η τρίτη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνδυάσουμε ε, τις δραστηριότητες και τα οικονομικά υπό καλές συνθήκες ε, που φυσικά είναι κάτι το Εγώ πιστεύω ότι τα οικονομικά όμως καθοδηγούν τις ε, δραστηριότητες και όχι το αντίστροφο. Πώς μπορούμε λοιπόν στον με τις εξυπηρέτησης να συνδυάσουμε όλα αυτά διότι μιλάμε για αυτό το one-stop shop πάντα, το γνωστό. Οπότε αυτό το one-stop shop αφορά περισσότερο τη γενική εξέλιξη των ε, των δραστηριοτήτων ή την οικονομική τους διαχείριση. Και τέλος, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, η παρουσίαση του κ. Σέκη μας έδειξε πολλά. Είδαμε δύο διαδρόμους σήμερα Είδαμε ένα διάδρομο των πλουσίων και των λιγότερο πλουσίων. Δεν το λέω για να δείξω ότι υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, αλλά βλέπετε τώρα. Ε, μόλις φύγουμε από τους πλούσιους τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα είναι περίπλοκες, ε, είναι πιο, πιο σύνθετες εργασίες ε, και γίνονται πιο απλές όπως καταβαίνουμε προς τα στα μέρη. Οπότε αυτό, τι γίνεται με τη γεωγραφική διαχείριση. Μπορείτε να εξηγήσετε λοιπόν σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ε, αυτό που λέμε ότι το σύνολο έχει μεγαλύτερη αξία από ότι τα επιμέρους κομμάτια του ε, τα κράτη-μέλη το καταλαβαίνουν αυτό και επίσης δεν θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε τους, θέσεις, τους ανθρώπους να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο από ότι τα επιμέρους κομμάτια. Και αυτή είναι η ερώτησή μου προς τους συντονιστές. Ε, αυτές οι οικονομικές διατησίε τελικά δεν γίνονται βάσει των πόσων χρημάτων μπορούν να δώσουν οι εταίροι. Ε, δηλαδή, όταν οι οικονομικοί εταίροι ε, χρηματοδοτούν το σύνολο ή ένα κομμάτι. Ε, και μια τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Σέκη. Τι γίνεται με τη συνδεση havris Χαύρις-Μανχάιμ που μου φαίνεται να ε, έχει ε, τεθεί στο πλάι, να το έχει καταλήψει το ενδιαφερόμενο κρατός μέλος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερικέ. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Σέκη, δεν καταλαβαίνω γιατί ο διάδρομος του Ατλαντικού σταματάει στο Παρίσι. Γιατί δεν πάει μέχρι το βορρά της Γαλλίας και το, περιοχή Νόρ Παντεκαλέ. Διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή θα ήταν λογικό ο, διάδρομος του Ατλαντικού να πάει μέχρι τον Νόρ Παντεκαλέ. Νορ Παντεκαλέ. Θα μου το εξηγήσετε. Και δεύτερον, μπορείτε να μου πείτε τι ρόλο έχετε εσείς ε, στη σχέση με τα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί κοιτώντας το διαδρόμο του Ατλαντικού, για πολύ καιρό υπήρξαν ε, διαφορές μεταξύ γαλλικής κυβέρνησης και ισπανικής κυβέρνησης ειδικότερα για αυτό το γνωστό, ε, τη γνωστό μεγάλη διαδρομή ε, συνδυοδρομική ε, και συστάθηκε μια ομάδα εργασία για να συντονίσει τι θέσει μεταξύ των χωρών κτλ. Εσεί ω συντονιστή συμμετείχατε σε αυτή την ομάδα εργασία και αν ναι, τι συμπεράσματα έχετε να μας παρουσιάσετε. και μετά μια ερώτηση για σας κύριε Κόξ. Υπάρχει αυτό το γνωστό τούνελ που μας λένε θα μας κοστίσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για να συνδέσει τη Σκανδιναβία με την Ήπειρο με την υπηρετική Ευρώπη. Και εγώ βλέπω το σύραγγα αυτή θα είναι μια σύραγγα υποβρύχια 18 χιλιόμετρων προς τη Δανία με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας και ήθελα να μου πείτε γιατί εδώ τίθεται το ζήτημα το κλιματικό και τη απαλλαγή από τι ανθρακούσε εκπομπέ. Είναι σημαντικό το διακύβευμα. Γιατί? Διότι οι κλιματικέ συνθήκε, ειδικότερα στη Βαλτική, μεταβάλλονται. Δεν είναι ίδιε με πριν από 10 χρόνια. Και πώ θα είναι άργε σε 10 ή 15 χρόνια η κατάσταση. Έχουν ληφθεί υπόψη αυτέ οι συνθήκε. Με τα ε, λέτε ότι θα γίνουν και άλλες οικονομίες πιστεύω ε, ε θα, τα φεριμπότ θα επηρεαστούν από όλο αυτό. Τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση. Και μετά μπορείτε να προβλέψετε κάτι όσον αφορά τις δαπάνες που δίνονται για αυτά τα προγράμματα αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος το οποίο δεν είναι αμεληταίο διότι είναι ένα κόστος σημαντικό. Αύριο δεν θα μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε τη φύση. Πώς θα γίνει να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ των διαφορών ε, παραγόντων. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σαντέρ για λίγα λεπτά, διότι θέλω οι συντονιστές μας να προλάβουν να απαντήσουν το σύνολο των ερωτήσεων. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε για ε, που, μου δίνει τον λόγο άργησα, είχαμε, ήμασταν στον δημοσιονομικό προπολογισμό, στην, ε, ε δημοσιονομικό έλεγχο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντονιστές και τον κύριο Σέγγι, και τον κύριο Κόξ που είναι συντονιστές οι οποίοι πραγματικά βοηθούν στο να προχωρήσουν όλα αυτά τα project ακόμα και πρώτο μεγαλύτερων δυσκολιών. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα αμυγός στον διάδρομο Ατλαντικού ε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σέκη, σε αυτήν την διακυβερνητική ομάδα Ισπανία, Πορτογαλία, Ισπανίας Πορτογαλίας, ε, η Πορτογαλία για πολιτικούς ε, λόγους αλλά και οικονομικούς ε, ήρθε μετά βέβαια, αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία υπάρχουν, το ΕΦΣΙ, το blending, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από πλευράς του Κοινοβουλίου, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα να μπορέσουν όντως να βοηθήσουν. Δεύτερον, θα ήθελα να ξέρω και ο κ. Κόξ και ο κ. Σέκη να μου πούν ποια είναι η άποψή τους, γι' αυτό προτείναμε ε, οι συντονιστές δηλαδή να λάβουν υπόψη τους στα διάφορα, στις διάφορες εκθέσεις τους πώς επηρεάζει τους διάφορους διαδρόμους και τις υποδομές ε, που χρηματοδοτούμε ε, για τη βελτίωση του switch, δηλαδή το πέρασμα ε, στο τρένο για τα εμπορεύματα, στις ρομικές μεταφορές και στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εσωτερικές πλουτές οδούς. Και τέλος για τους ισπανικούς λιμένες υπήρχε μια ερμηνεία κάπως sui generis για την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου τον κύριο κάμπ να πω αφενός ε, ότι αυτή η έκθεση ε, προέκυψε τη στιγμή της μεγάλης κρίσης ε, της Ισπανίας. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ανάπτυξη και ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η επίθεση είναι επειδή υπάρχει ο φόβος ε, τα ισπανικά λιμάνια να είναι πιο ανταγωνιστικά από το Ρότερνταμ. Ε, αυτά τα μεγάλα λιμάνια θα έχουν τελικά μέλλον. Να ευχαριστώ στο λόγο τώρα στους συντονιστές για να απαντήσουν στα ερωτήματα. Στις 12.30 όμως πρέπει να φύγουμε από την αίθουσα, οπότε πέντε λεπτά ο καθένας για να δώσει τόσο γίνεται περισσότερες απαντήσεις. Θα πάω γρήγορα, όπως τα τρένα, τα σημερινά και τα αυριανά. Ο κύριος Έρτου μίλησε για το μοντέλο που έχουμε. Νομίζω ότι είναι μοναδικό και αποτελεσματικό. Είναι ένα μοντέλο συνεργασίας, διαλόγου και δημιουργικότητας. Πρόκειται για μια εταιρική σχέση η οποία ε, ε, πηγαίνει και από τα πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω προς τα πάνω. Περιλαμβάνει ομολόγους ε, και ομότιμους και νομίζω ότι είναι το καλύτερο μοντέλο διακυβέρνησης και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα προσμίμησης για πάρα, προσμίμησης για πάρα πολλούς άλλους τομείς. Ο κύριος Βάντεκα μίλησε για στεγανά, μα γι' αυτό ακριβώς κάνουμε. Ε, αυτή την, ε, τη διαδικασία ακριβώς για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Πολλοί συνάδελφοι ε, μίλησαν για τους χώρους πρόσβασης, ιδίως για τον Μπρένερ. Δεν είναι σωστό να πούμε ότι η Ιταλία έχει μείνει, έχει μείνει πίσω. Ίσα ίσα 13 χιλιόμετρα έχει δεσμευτεί η Ιταλία να ολοκληρώσει στον νότιο άξονα του διαδρόμου. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά, μάλιστα στο να επιτύχουμε τη συγχρηματοδότηση. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ θετικά τα νέα αυτά και η Ιταλία έχει δεσμευτεί ότι θα, θα προχωρήσει στο έργο. Για τη βόρεια πρόσβαση στον στο Μπρένερ, εκεί πράγματι υπάρχει ένα θέμα με τη χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά έχουν ε, σημειωθεί, έχει σημειωθεί ε, τους τελευταίους 12 μήνες. Για το ΑΕ που είπε η κυρία Μάισνερ, ναι, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε, ε, ε, είναι μία από τις προτεραιότητες ε, του Ομοσπονδιακού Σχεδίου για τα οδικά δέκτυα. Το εκτιμόμενο κόστος είναι 3,8 δισεκατομμύρια έργα, ε, η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι το 2030. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία προκειμένου να ε, εξευρεθεί χρηματοδότηση αλλά και να προχωρήσουν τα σχέδια αυτοματοποίησης του έργου. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα και τα άλλα ζητήματα που ρωτήσατε, στο σχέδιο 3 του διαδρόμου που επεξεργαζόμαστε τώρα ε, αρχίζουμε και ασχολούμαστε σε βάθος με αυτά τα ζητήματα γιατί μέχρι στιγμής ε, ε, γνωρίζαμε ποιος είναι ο διάδρομος και πού είναι οι ελλείψεις, τα χάσματα. παρόλα αυτά τώρα πια είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε και με αυτά τα ζητήματα και θα είμαστε σε επαφή για να σας ενημερώνω αν θέλετε τα επόμενα δύο χρόνια καθώς θα δίνονται απαντήσεις. Ε, ε, η κυρία Κλούν μίλησε για την ε, διασύνδεση και τα σχετικά ζητήματα της περιφέρειας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στις επισκέψεις μας στο, στα, στα λιμάνια ε, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τις αρχές, ε, βρισκόμαστε σε επαφή με την Επιτροπή, με όλες τις αρμόδιες αρχές, ε, διοργανώνουμε σεμινάρια. Υπάρχει λοιπόν ένας υψηλού επίπεδου συντονισμός για την, περιφά... την περιφέρεια. Εγώ πιστεύω πολύ στην ισότητα που κατοχυρώνεται μεταξύ των κρατών μελών στις συνθήκες. Για το ζήτημα λοιπόν της, της περιφέρειας, αν ο κόλπος του Μπότνια μπορεί να ενταχθεί, εμείς δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και σχετικές πρωτοβουλίες ε, οι τοπικές αρχές ε, της Στοκχόλμης και του Γκέτεμπορκ για τη στρατηγική Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε επ' αυτής και νομίζω ότι το ITS δεν πρέπει να περιοριστεί σε στεγανά. Πρέπει να ε, αποτελέσει ένα, μια από τις βασικές διαστάσεις που θα λαμβάνονται υπόψη καθολικά στην, ε, στο σχεδιασμό των έργων μας. Κύριε Ρικέ, νομίζω ότι τα ερωτήματά σας είχαν ε, πιο οικονομικό χαρακτήρα αφορούσαν τη χρηματοδότηση. Θα σας απαντήσει ο κύριος Σέκη. Να πω επίσης ότι η διασύνδεση Φέλμαν ε, θεωρούμε ότι θα αποσυμφορήσει ε, σε σημαντικό βαθμό τις εμπορευματικές ροές από άλλους τρόπους μεταφοράς ε, νομίζω ότι ε, αυτή τη στιγμή η, ο μεγαλύτερος όγκος ε, πραγματικά μεταφορών γίνεται μέσω ε, πλοίων, ε, πορθμίων και φορτηγών. Αυτό θα αλλάξει με, τον, με, τα, με το νέο έργο και αυτό, προς αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, προκειμένου πραγματικά να αξιοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ε, μακροπρόθεσμα. Άρα, από αυτή την άποψη, οι προσδοκίες μας είναι θετικές. Αυτά, νομίζω εγώ, είχα να πω. Ευχαριστώ, ο κύριος Σέκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ήταν όλα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια βέβαια ήταν πολύ λεπτομερή, οπότε θα μπορούσαμε και με διμερή επαφή να σας απαντήσω σε αυτήν. Ο κύριος Έρτουγκ ρώτησε για τις κυβερνήσεις και την εμπλοκή τους. Ε, οι δικές μου εμπειρίες είναι πραγματικά πολύ θετικές. Ε, ιδίως στην περιοχή Μάνχαιμ Στρασβούργου που επικαλύπτεται και με τον διάδρομο ε, Σκανδιναβίας Μεσογείου έχουμε μάλιστα προχωρήσει και σε κοινέ δράσεις ε, που αφορούν τις εσωτερικές πλωτές οδούς τις ε, ε σχέσεις μεταξύ τοπικών κοινοτήτων στις διασυνοριακές περιοχές για, το, για το ζητήματα των εμπορευματικών μεταφορών στο Μάνχαιμ υποβάλλονται προτάσεις έργων. Βεβαίως θα χρειαστεί χρόνος για να τεθούν υπο, σε επεξεργασία και να αξιολογηθούν, αλλά είναι και αυτό ένα τμήμα της κοινή μας προσοχής που δίνουμε για την προώθηση. Οι διάδρομοι ακολουθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τουλάχιστον από δύο απόψεις. Όχι μόνο, ε, δεν είναι μόνο το ζήτημα των διαφορετικών οδικών δικτύων και των διαφορετικών υποδομών, αλλά ε, αφορούν και ε, πιο οριζόντια ζητήματα, ITS, καθαρή ενέργεια κτλ. Και, Και καθώς καταρτίζουμε τα σχέδια εργασιών μας, προσπαθούμε όλο και περισσότερο να ακολουθούμε μια τέτοια ενιαία, ολοκληρωμένη προσέγγιση και να λειτουργεί ο διάδρομος ως μια μήτρα κατά κάποιο τρόπο και όχι ως ε, ένας κατάλογος διαφόρων έργων που πρόκειται να συνδεθούν. Οι διάδρομοι έχουν πραγματικά αυτό που αποκαλούμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και γι' αυτό και χρειάζεται χρηματοδότηση που θα αφορά όχι μόνο την ποιότητα ε, του, του έργου αλλά και της ευρωπαϊκής προσδεχόμενης αξίας, της δασυνορικότητας κτλ. Ενιά θηρίδα. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να μειώσουμε την γραφειοκρατία που χρειάζεται κανείς να, να περάσει με, με, έως ότου πάρει το πράσινο φως για την, ολοκλήρωση, για την ε, κατασκευή ενός έργου. Όλο και περισσότερο το One Stop Shop είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ασχολείται με την υλοποίηση του ΕΦΣΥ και που στο μέλλον θα εμπλέκεται όλο και περισσότερο ε, στις μεικτές ε, δραστηριότητες η Ισλανδία είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι κομμάτι του διαδρόμου, αλλά εμείς ε, τους έχουμε στο νου μας. Ε, ε, το ίδιο και με, όσον αφορά την Πορτογαλία και την Ισπανία φυσικά. Και για τη μελλοντική αναθεώρηση θα ψάξουμε να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ε, όταν θα ονομάζουμε ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο core ε, πυρήνα, θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι ενός δικτύου. Τα ομόλογα έργων ήταν μια πολύ καλή ιδέα πριν 5-6 χρόνια. Τα project bonds αυτά, τα ομόλογα έργων, έχουν μετασχηματιστεί σε εργαλεία εγγυητικά ονομάζονταν project bonds της Κομισιόν ε, στην προηγούμενη περίοδο και ήταν η, προ... η πρόδρομη του ΕΦΣΙ ουσιαστικά. Αυτό μελετά το ΕΦΣΙ, τι είναι δυνατόν να γίνει με αυτά. Και σήμερα ανήκουν στην αμυκτή προσέγγιση, ε, σημαντική συνιστόσα της οποίας είναι το ΕΦΣΙ. Στο μεταξύ, για να κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα, χρησιμοποιούμε για τα bonds αυτά, για τα ομόλογα αυτά που μπαίνουν στην αγορά για μια συγκεκριμένη περίοδο, για συγκεκριμένα έργο όπως για το λιμάνι του Καλέ ε, και μετά έχουμε τις μακροχρόνιες επενδύσεις. που συνδυάζονται με αυτά τα ομόλογα. Λοιπόν, η ιδέα μας είναι να συντεριάξουμε δηλαδή τη μακροχρόνια διάσταση απόψης ζήτησης αλλά και από την άποψη της χρηματοδότησης ε, με τον καλύτερο θεσμικό τρόπο. Αυτό υλοποιείται αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, πώς λειτουργεί το πιλωτάζ, διαχείριση. Τι μπορώ να σας πω στην παρουσιαφάση... βρισκόμαστε σε εργαστηριακή φάση. Το blending call είναι η νέα πρόκληση και θα προκαλέσει πιστεύουμε το ενδιαφέρον ε, των δικαιούχων. Πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα μας δώσει και κάποια εμπειρία. και στην επόμενη οικονομική περίοδο θα δημιουργήσουμε βάσει αυτής της εμπειρίας ένα νέο εργαλείο. Δεν λέω ότι κάνουμε τα πάντα προσαρμοσμένα κατά περίπτωση, αλλά το τι θα γίνει στην πρακτική μέχρι τον Ιούλιο, που είναι η προθεσμία για το πρώτο κομμάτι και μετά στη δεύτερη φάση, Ιούλιο από τη στιγμή που θα υπογραφεί οριστικά και θα δοθούν τα χρήματα, θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Η μέθοδος είναι σαφής, η ιδέα είναι σαφής, τις λεπτομέρειες θα προσπαθήσουμε να τις καταλάβουμε μαζί με τους δικαιούχους της προσέγγισης αυτής. Merci Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τους συντονιστές για τις παρουσιάσεις αυτές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, ελπίζω. Πάντως ολοκληρώνεται τώρα η συνεδρίασή μας. Θα σας στείλουμε mail όποια άλλα στοιχεία προκύψουν. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρίασή μας. Να σας πω ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 10 ε, Απριλίου στις 3. Σας ευχαριστώ όλους.